Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διατάξη προβλέπει τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την κατάσταση στην Πολωνία. Κυρίες και κύριοι σας, επισημαίνω ότι σε αυτό το κομμάτι των συζητήσεων δεν προβλέπεται διαδικασία catch the eye και δεν θα επιτραπούν μπλε κάρτες. Όχι, δεν αφήνουμε να γίνει συζήτηση επί του κανονισμού. Ξεκινούμε τη συζήτησή μας. Το αποφάσισε η διάσκεψη των Προέδρων και έχει ενημερωθεί κάθε πολιτική ομάδα. Κυρία Πρωθυπουργέ, κυρία Σίτλου, καθώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίες και κύριοι, η απόφαση για τα μέτρα που σκοπεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εκκίνηση διαλόγου σχετικά με την κατάσταση στην Πολωνία και την αξιολόγηση με όρους του πλαισίου για το κράτος δικαίου αποτελούν ε, μια πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα νέο μέσο, ένα νέο μέτρο που μέχρι τώρα δεν έχει ε, χρησιμοποιηθεί παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το Μάρτιο του 2014 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως μηχανισμός έγκαιρης προειδοποίησης. Το κράτος δικαίου ξέρουμε τι συνεπάγεται. Διάκριση εξουσιών και δεν είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα, αλλά όρο διαφύλαξης της δημοκρατίας και των κοινωνικών μας μοντέλων. Άρα πρόκειται για μια συζήτηση κεντρικής σημασίας για το μέλλον. Και θεωρώ ως εκ τούτου ότι η συζήτηση θα γίνει με τρόπο συντονισμένο, συγκεντρωμένο και σεβασμό του ενός προς τον άλλον. Καλώς ήρθατε λοιπόν για άλλη μια φορά κυρία Πρωθυπουργέ. Ευχαριστώ βεβαίως για την αποδοχή της πρόσκλησης συμμετοχή στη συζήτηση. Προχωρώ στη συζήτηση. Εξ ονόματος του Συμβουλίου και εκπροσωπών την Προεδρία, ο κύριος Κέντερς από τις κάτω χώρες. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο μια αγορά, είναι και μια ένωση που έχει χτιστεί πάνω σε κοινέ αξίες. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες είναι ξεκάθαρες. Τα διάφορα άρθρα αναφέρουν τις αξίες πάνω στις οποίες έχει χτιστεί αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και φροντίζει εξή αυτές να είναι κοινέ μεταξύ όλων μας. Το να ανήκει κανεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σημαίνει μόνο ωφέλη, σημαίνει και υποχρεώσει. Και μια από τι κύριε υποχρεώσει τη κάθε χώρα μέλη είναι να σέβεται τι θεμελιώδεις αξίες τη Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίω το κράτο δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι ακριβώ αυτό που μα κάνει χώρε μέλη, αλλά είναι και αυτό που κάνει την Ευρωπαϊκή Ένωση μοναδική στον κόσμο. Και είναι αξίε που μοιραζόμαστε μεταξύ μα, όχι μόνο γιατί είναι γραμμένε κάπου, αλλά γιατί έχουν πάρει ζωή στις ανοιχτές μας κοινωνίες τις τελευταίες δεκαετίες. Μερικές φορές ξέρουμε ότι είναι θεμελιώδεις επειδή διασφαλίζουν την ελευθερία των πολιτών μας και τη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Όμως, ούτε το κράτος δικαίου, ούτε καμιά άλλη θεμελιώδης αξία δεν είναι από μόνη της κάτι το αυτονόητο. Και αυτό το ξέρουμε μέσα από το δογματισμό που έχουμε δει πολλές φορές. Έχουμε πάρει τα μαθήματά μας και τα έχουμε πάρει με το χειρότερο τρόπο. Και πολλές φορές έχουμε υποσχεθεί στους εαυτούς μας ότι δεν θα γυρίσουμε σε εκείνες τις σκοτεινές εποχές, ότι θα φτιάξουμε μια νέα κοινότητα όπου θα κυριαρχεί η ελευθερία και η δημοκρατία. Και το πετύχαμε. Και το μυστικό της επιτυχίας αυτής είναι ότι βάλαμε τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου πάνω απ' όλα. Και παραμένει και σήμερα ζωτική σημασία να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια είναι μια συνεχής πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι κυβερνήσεις των χωρών μα, αλλά είμαστε ειλικρινεί. Δεν υπάρχει καμία χώρα που έχει το μονοπόλιο της αρετής και καμία χώρα δεν έχει και το μονοπόλιο του κακού. Όλοι έχουμε αδυναμίε. όμως η δύναμη των δημοκρατιών μας είναι ακριβώς ότι μπορούμε τις αδυναμίες αυτέ να τι εντοπίσουμε και να τις αναγνωρίσουμε και να τις διορθώσουμε στη συνέχεια. Αυτό είναι η δημοκρατία. Αυτό σημαίνει επίση ότι είμαστε έτοιμοι να έχουμε ανοιχτέ συζητήσει μεταξύ μα για τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προστατεύσουμε τι αξίε και τι αρχέ αυτέ. Η σημερινή συζήτηση λοιπόν, όπου κλήθηκε να παρεύει και το Συμβούλιο και σα ευχαριστώ αυτό, απορρέει από τα πρόσφατα μέτρα που εισήγαγε η νεοεκλεγμένη κυβέρνηση στην Πολωνία. Τα μέτρα αυτά κυρίως οι θέσεις του συνταγματικού δικαστηρίου και οι θέσεις στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα μας έκαναν να έρθουμε εδώ σήμερα και να συζητήσουμε. Όντως το κράτος δικαίου είναι κάτι που πρέπει να υπερισχύει σε κάθε χώρα. Η ελευθερία λοιπόν λόγου, η ελευθερία, ο πλουραλισμός στα μέσα ενημέρωσης αποτελούν και τον ακρογωνίο λίθο για την δημοκρατία μας. Πρέπει να δούμε λοιπόν ποιες είναι οι επιπτώσεις στην κοινή γνώμη και πώς έχει συμμετοχή των πολιτών. Πολλές φορές το Συμβούλιο μέχρι σήμερα έχει υπογραμμίσει ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη η δικαιοσύνη και ότι αυτή είναι μια πολύ βασική αξία που απορρέει από τις δημοτικές παραδόσεις των χωρών μελών. Δεν είναι βέβαια η Προεδρία η οποία θα κρίνει. Το Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει αυτή την υπόθεση. Θέλω όμως σύντομα να πω δύο λόγια για την Πολωνία. Αρκετές χώρες έχουν υποφέρει τα τελευταία χρόνια, αλλά η Πολωνία πολύ περισσότερο τις δεκαετίες που έχουν περάσει. Αλλά το πνεύμα της Πολωνίας δεν έχει πεθάνει. Παρέμεινε ζωντανό, ακόμα και κάτω από το ρωσικό ζυγό και βοήθησαν πολωνικά στρατεύματα να απελευθερωθεί και δικιά μου χώρα. Γι' αυτό και είμαι ευγνώμων στην Πολωνία. Τώρα είμαστε στο 2016. 11 χρόνια είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Πολωνία. Και σήμερα βρίσκεται στον κύκλο των μεγάλων δυνάμεων. Κατάφερε να γίνει μια δύναμη επιτυχημένη οικονομικά και κοινωνικά και να ενισχύσει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Οι Πολωνοί τα κατάφεραν γιατί βασίστηκαν στην παράδοσή τους και επειδή έχουν ένα από τα πιο πεφωτισμένα συντάγματα οι Πολωνοί λοιπόν αξίζουν κάθε σεβασμό για τόσα έχουν πετύχει. Ζητούν κυριαρχία, εθνική κυριαρχία και γι' αυτό ακριβώς βρίσκονται και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προεδρία είναι ευγνώμων λοιπόν που τη δώσατε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε αυτή τη συζήτηση και το κοινοβούλιο σα πάντα έδειξε την αφοσίωσή του στο κράτο δικαίου, τη δημοκρατία και τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι μυστικό ότι η χώρα μου, οι κάτω χώρε που φιλοξενεί διάφορα διεθνή δικαστήρια, θεωρεί πολύ σημαντικά τα θεμελιώδη δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Το 2013 με την Γερμανία, τη Φιλανδία και τη Δανία στείλαμε επιστολή στους εταίρους μας για να πούμε ότι χρειάζεται μια πλατφόρμα για να συζητιώνται τα θέματα του κράτους δικαίου. Αφού μιλάμε για οικονομικά ζητήματα, γιατί να μην μιλήσουμε και για το κράτο δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό και οργανώνουμε ένα σεμινάριο στο Στρασβούρο στι 2 Φεβρουαρίου για τη μετανάστευση και το κράτο δικαίου. Και ελπίζω να έρθουν πολλοί συμμετέχοντε. Πριν από δύο μήνε το Συμβούλιο ξεκίνησε το διάλογο για το κράτο δικαίου στην Ένωση. Θα οργανώσουμε και ένα δεύτερο διάλογο κάποια στιγμή τον Μάιο και θα χρησιμοποιήσουμε τα αποτελέσματα του σεμιναρίου του Φεβρουαρίου στη συζήτηση ακριβώ αυτή θέλουμε να σεβόμαστε τις βασικές μας αξίες. Βέβαια το Συμβούλιο δεν είναι μόνο του στα θέματα αυτά που έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Αντίθετα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη γνώμη μας έχει σημαντικό ρόλο να παίξει σε αυτόν τον τομέα. Ακριβώς επειδή είναι και ο θεματοφύλακας των συνθηκών. Θέλω εδώ να τονίσω και τον ρόλο του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Επιτροπής της Βενετίας για αυτά τα ζητήματα. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επιτροπή της Βενετίας εξετάζουν τις εξελίξεις και θα παρακολουθήσουν τη σημερινή συζήτηση. Γι' αυτό και προτείνω η σημερινή συζήτηση να γίνει αμερόληπτα, με πνεύμα συνεργασίας μεταξύ μας και να καταλήξουμε σε πρόοδο αφού έχουμε αναλύσει τα γεγονότα. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα να μας ενημερώσει για τις εργασίες της Επιτροπής μετά την συνεδρία της προηγούμενης εβδομάδας και τις συζητήσεις με τις πολωνικές αρχές. Και η Πρωθυπουργό Σίτλο, με την οποία είχα την τιμή να συζητήσω σήμερα, θα πάρει το λόγο εδώ και θα παρουσιάσει τη δικιά της θέση. Η συμμετοχή όλων σήμερα θα συνεισφέρει σε ένα διάλογο μέσα στην ευρωπαϊκή μας δημοκρατία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής. Κυρίες και κύριοι, στα θεωρία προσκεκλημένοι μας, καλώς ήρθατε, είστε πολλοί, έχετε ταξιδέψει από μακρινές αποστάσεις. Σας επισημαίνω ωστόσο ότι ο κανονισμός λειτουργίας του Κοινοβουλίου δεν επιτρέπει ε, χειροκροτήματα ή αποδοκιμασίας από την από τα θεωρία και σας καλώ να, να διατηρήσετε την ιδιαιτερότητά σας να παρακολουθείτε τη συζήτηση. Ο κύριος Τίμερμαν, ως πρόεδρος, της, αντιπρόεδρος Επιτροπής. Κύριε Πρόεδρε του Κοινοβουλίου, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίε και κύριοι το μέλη του Κοινοβουλίου. Εκ μέρου των συναδέλφων μου τη Επιτροπή και μου του Ιδίου, θέλω να σα δώσω του λόγου για του οποίου αποφάσισα να αξιολογήσει τα πρόσφατα γεγονότα στην Πολωνία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πώ σκοπεύουμε να προχωρήσουμε με επικοδομητικό τρόπο και να έχουμε διάλογο βασισμένο στα γεγονότα με την Πολωνία για να αποφύγουμε την ανάδυση ενό ε, συστηματικού κινδύνου κατά του ε, κράτου δικαίου. Ο βασικό λόγο που θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία αξιολόγηση βάσει του πλαισίου δικαίου του 2014 θα είναι, είναι οι πρόσφατες αποφάσεις για το συνταγματικό δικαστήριο και η διαφωνία για τον αριθμό δικαστών που συμμετέχουν στο δικαστήριο αυτό επί της αρχής. Αυτό το ζήτημα θα πρέπει να το λύσει το συνταγματικό δικαστήριο το ίδιο. Ωστόσο, όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, τα άλλα θεσμικά όργανα του πολωνικού κράτους δεν έχουν συμμορφωθεί με τις αποφάσεις του συνταγματικού δικαστηρίου επί του θέματος. Αυτό έχει δώσει λαβή για να ε, εκφραστούν αβεβαιότητες για την ε, ίδια τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου στην ε, Πολωνία. Επιπλέον, το Πολωνικό Κοινοβούλιο αποφάσισε να συντομεύσει τη θητεία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δικαστηρίου στις 28 Δεκεμβρίου του 2015 μια τροπολογία για το νομοσχέδιο και το ιδιωτικό καταστατικό του ε, Συνταγματικού Δικαστηρίου άρχισε να ισχύει και δίνει την εντύπωση ότι η λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου θα δυσχεραθεί ιδιαίτερος δεδομένης της ε, κέρια σημασίας του συνταγματικού δικαστηρίου για το σύνολο του πολωνικού δικαστικού συστήματος, φοβούμαστε ότι θα αναδυθεί ένα συστημικός κίνδυνος εις βάρος του κράτους δικαίου στη χώρα. Επίσης, εκφράστηκαν ανησυχίες σε ό,τι αφορά το, νέο νόμο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το κράτος δικαίου, όπως ορίζεται στο πλαίσιο μας για το κράτος δικαίου, απαιτεί την, τον σεβασμό της δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης και η πολυφωνία συνδέονται στενά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Όλος ιδιαίτερος με την ελευθερία της έκφρασης. Γι' αυτόν τον λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί αναγκαίο να αποτιμήσει τον νόμο αυτό υπό το φως του συγκεκριμένου πλαισίου που διαθέτουμε για το κράτος δικαίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεμελιωθεί σε ένα κοινό σύνολο αξιών όπως εκφράζονται στο άρθρο 2 για την ε, συνθήκη, από, τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάνει ιδιαίτερη μνήα για το σεβασμό του κάτω δικαίου. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ε, νομικών του συστημάτων εξαρτάται από την εμπιστοσύνη και την πίστη ότι το κάτω δικαίου τηρείται με τον ίδιο αυστηρό τρόπο σε όλα τα κράτη-μέλη. Όταν ε, οι εθνικές διασφαλίσεις για το κάτω δικαίου φαίνεται να απειλούνται, τότε η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναλάβει δράση. Επίσης, να σημειώσω ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Πολωνία έχει κύριο ρόλο να διαδραματίσει, προκειμένου και οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που τώρα προγραμματίζονται στην Πολωνία θα συμμορφώνονται και θα συνάδουν με το Σύνταγμα. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι καθοριστική σημασία η σημερινή αντιπαράθεση σε ό,τι αφορά το Συνταγματικό Δικαστήριο της Πολωνίας να επιληθεί κατεπηγόντως, ώστε το δικαστήριο να διαδραματίσει το ρόλο του ως ένας μηχανισμός που συμμετέχει στο εθνικό σύστημα κράτους δικαίου. Απίθυνε επιστολή δι προ την Πολωνία στι 23 και 30 Δεκεμβρίου του 2015 για το θέμα αυτό, όμω οι απαντήσει που λάβαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκτοτε δεν ήταν πλήρε, ήταν ανεπαρκεί ώστε να διασκεδάσουν τι ανησυχίε μα. Το πλαίσιο του κράτους δικαίου επιτρέπει να αποτιμήσουμε το όλο θέμα με έναν τρόπο διαρθρωμένο σε ένα διάλογο με τις πολωνικές αρχές. Θα έπρεπε λοιπόν να αξιοποιήσουμε το πλαίσιο κράτους δικαίου με έναν τρόπο δημοκρατικό και επικοδομητικό, σε ένα πνεύμα συνεργασίας και όχι αντιπαράθεσης. Είδαμε ε, ότι προ λίγου... Ε, ε, στην επιστολή μου της περασμένης εβδομάδας μόλις μου απευθύνθηκε μία απάντηση, μία επιστολή. Θα την αναλύσουμε λοιπόν για να δούμε κατά πόσον οι ερωτήσεις που απευθύναμε την περασμένη εβδομάδα είναι επαρκείς αυτή τη στιγμή. Φυσικά δεν μπορώ να πω τώρα σε λεπτομέρειες γιατί πρέπει να το εξετάσουν ε, οι συνεργάτες μου και την επιστολή λάβαμε μόλις πριν από μία ώρα περίπου. Να τονίσω ότι βρισκόμαστε στην έναρξη της διαδικασίας που προβλέπει το πλαίσιο. Το πλαίσιο έχει χαρακτήρα προληπτικό και το να επικεντρωθούμε στα αντικειμενικά, νομικά και σε σχέση με τα γεγονότα στοιχεία δεν σημαίνει ότι προδικάζουμε τις επόμενες φάσεις της διαδικασίας. Θα βασιστούν όλα στα γεγονότα που υπάρχουν και στις απαντήσεις που θα λάβουμε. Ο διάλογος μπορεί να είναι και έντονος και να καταλήξει πολύ γρήγορα σε όριμα αποτελέσματα. Η συμμετοχή στο διάλογο θα είναι αμερόληπτη, θα βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία και θα γίνει σε πνεύμα συνεργασίας. Είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σέβεται την ε, κυριαρχία της Δημοκρατίας της Πολωνίας και θα ασκήσει τα καθήκοντά της με τρόπο αντικειμενικό και χωρίς καμία παρεμβατική τάση, όπως και για άλλα κράτη-μέλη, βάσει των ε, υποχρεώσεων που προβλέπονται για την Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τι συνθήκε που έχουν υπογράψει και κυρώσει τα κυρίαρχα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, τέλος, θα ολοκληρώσουμε θα διεξεγάγουμε μάλλον την ε, αποτίμησή μα αυτή σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Καλωσορίζω το γεγονό αυτό μετά την προτροπή μου προ την πολωνική κυβέρνηση, καθώ και εκείνη ζήτησε την γνωμοδότηση τη αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου για τη μεταρρύθμιση τη λειτουργία του Συνταγματικού Δικαστηρίου. Σε αυτό το πλαίσιο απευθύναμε επιστολή προ την πολωνική κυβέρνηση μόλι την περασμένη εβδομάδα. Έχω την αίσθηση ότι σε αυτό το πνεύμα ε, μα απίφθινε και απάντηση η πολωνική κυβέρνηση στην επιστολή τη της εβδομάδας. Θα αναλύσουμε προσεκτικά την απάντηση αυτή για τα περαιτέρω στάδια διαλόγου με την πολωνική κυβέρνηση, ελπίζοντας ότι το ζήτημα θα επιληθεί πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Τίμερμαντ. Το λόγο τώρα έχει η Πρωθυπουργός της Πολωνίας, κυρία Σίγκλου. Κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, και κύριοι. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να πω δύο λόγια για την Πολωνία σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω ότι η συζήτηση θα δεξαχθεί επί της ουσίας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για μένα για να μπορέσω να διασκεδάσω αμφιβολίε ή ανησυχίε που ενδεχομένω έχετε ακόμη ως προς την νομοθεσία που εισάγουμε, τις αλλαγέ που εισάγουμε στην Πολωνία αυτή τη στιγμή και γιατί το πράττουμε. Ύστερα από τις ε, εκλογέ του Οκτωβρίου, οι Πολωνοί πολίτες, αποφασίζοντα δημοκρατικά, επέλεξαν να εκδηλώσουν την προτίμησή τους προς τις αλλαγές αυτές τις οποίες είχε προτείνει η δική μου πολιτική οικογένεια, το δικό μου πολιτικό κόμμα, το κόμμα Δίκαιο και Δικαιοσύνη. Αυτή ήταν η επιλογή τους. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω σήμερα, ο οποίος σας εξ ε, του ευρωπαϊκού, του πολωνικού λαού. Βεβαίως, το δίκαιο το κράτος δικαίου είναι απαράβατα σε αξίες. Είναι αξίες και δικαιώματα για τα οποία αγωνίστηκαν οι Πολωνοί για πολλά χρόνια και έχουν στη σημασία για μας. Η ελευθερία, η εθνική κυριαρχία, η δικαιοσύνη. Είναι οι αξίες που μας καθοδηγούν στο έργο για την ανάπτυξη της χώρας μας. και ελπίζω ειλικρινά ότι μετά τη σημερινή μου αγόρευση θα πιστείτε πως η Ευρώπη, πως η Πολωνία ανήκει στην Ενωμένη Ευρώπη όπως ακριβώς ανήκουν και τα άλλα κράτη, τα κράτη που εσείς εκπροσωπείτε στο σώμα. Κυρίες και κύριοι, ακούμε, ακούμε να υψώνονται φωνές στην Πολωνία, φωνές που μας λυπούν, που είναι άδικες πολλές φορές, που κρίνουν και κατακρίνουν την πολωνική κυβέρνηση, κατά τρόπο άδικο. Αυτές οι άδικες φωνές ελπίζω ότι προκύπτουν μόνο από παρεξηγήσεις, από ανεπαρκή πληροφόρηση και ότι δεν είναι φωνές που καθοδηγούν οι κακές προθέσεις ή ότι αυτές είναι μόνο μειονότητα. Εμείς ως Πολωνοί οφείλουμε να προχωρήσουμε σε αυτό το κοινό εγχείρημα στηριζόμενοι στην διαφορά μας. Στο πλαίσιο αυτής της διαφοράς θέλουμε να οικοδομήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η πρόκληση. Γιατί οι αξίες της δικαιοσύνης είναι πολύτιμες για μας, όπως άλλωστε και της ενότητας, γιατί μια Ευρώπη ενωμένη, μια Ευρώπη ισχυρή ως δεσμίδα των ισχυρών κρατών μπορεί να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις. Και στο όνομα αυτών των μεγάλων προκλήσεων πρέπει να είμαστε σε θέση να μιλάμε ειλικρινά, να κοιτάμε ένα τον άλλο στα μάτια. Οι Πολωνοί λοιπόν θέλουν να στηρίξουν στις δύσκολες αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε διατεθειμένοι και θέλουμε να στηρίξουμε την Ευρώπη όταν καλείται να έρθει το με τις μεγάλες προκλήσεις. Είναι αξία αδιαπραγμάτευτη για μας η Ευρώπη. Και κύριε Υπουργέ, η ιστορία μας, και σας ευχαριστώ για τα λόγια που αφιερώσατε σε μας, η ιστορία μας είναι μια ιστορία δύσκολη, μια ιστορία που μας έφτασε μέχρι τη σημερινή εποχή, μια ιστορία γραμμένη με το αίμα που έχησαν οι γονείς και οι παππούδες μας που μας επιτρέπει σήμερα να ανήκουμε σε αυτή την Ενωμένη Ευρώπη. Οι άνθρωποι αυτοί έχησαν το αίμα τους και για άλλες χώρες της Ευρώπης και για άλλα έθνη. Αγωνιστήκαμε λοιπόν για χρόνια για να μπορούμε να εκφράζουμε ελεύθερα την ε, βούλησή μας, ε, τη σκέψη μας, να χτίσουμε το κράτος μας τα καταφέραμε. Δεν θα επιτρέψουμε να μας στερήσει κανείς αυτό το δικαίωμα γιατί για μας αυτή είναι η κοινή Ευρώπη. Είμαστε Ευρωπαίοι και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Οι Πολωνοί με τις ε, εκλογές του τελευταίου πόρου υποστήριξαν ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα του κόμματός μας, του κόμματος Δίκαιο και Δικαιοσύνη, το πρόγραμμα της κυβέρνησής μας ένα πρόγραμμα που απευθύνεται πάνω απ' όλα σε εκείνους άντρες και γυναίκες που σήμερα, ύστερα από τόσα χρόνια μετάλλαξης, αλλαγής και συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη ζωή τους. Ίσως αυτό σας ξαφνιάσει. Αλλά θα σας πω ότι η Πολωνία, μεγάλο κράτος και μέλος σημαντικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει σημαντικά προβλήματα, όπως πολύ ψηλή ανεργία των νέων, αβεβές ε, συνθήκες εργασίας για τους νέους, παιδιά τα οποία ελπίζουν να πάνε στο σχολείο για να φάνε το μόνο ζεστό γεύμα της ημέρας. Ε, ηλικιωμένους που πρέπει να διαθέσουν τη μισή του σύνταξη για τα φάρμακά τους, που συχνά βρισκόνται ενώπιον του σκληρού διλήμματος να αγοράσουν φάρμακα ή να πληρώσουν το λογαριασμό του ηλεκτρικού. Αυτό αντιμετωπίζουν πολλοί Πολωνοί. Και πολλοί Πολωνοί έχουν ε, την αίσθηση ότι τους ε, ξέχασαν σε αυτή τη διαδικασία της μεταλλαγής της χώρας, ότι λησμονήθηκαν. Και τώρα έχουμε μια Πολωνία κράτος ευρωπαϊκό, ε, μια Πολωνία των ίσων ευκαιριών, των ελευθεριών, που θέλουμε να προσφέρουμε στον ίδιο βαθμό προς όλους. Έχουμε προτείνει λύσεις που έχουν αποδώσει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εμπνεόμενοι από τις βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών και είμαστε πεπισμένοι ότι αυτό οφείλαμε να κάνουμε, να μιμηθούμε αυτούς που έχουν επιτύχει και μπορούν να δείξουν το δρόμο. Ταυτόχρονα βλέπουμε ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες έχουν την εντύπωση πως πρέπει να εξασφαλιστούν οι συνθήκες ίσης ευκαιρίας για το καθένα. Σε αυτό ακριβώς, σε αυτή τη θεωρία στηρίζεται το πρόγραμμα μας για την Πολωνία. Οι εκλογές αυτές που οδήγησαν στην ε, στο σχηματισμό της κυβέρνησης, οι επιλογές αυτές του πολωνικού λαού μας οδήγησαν στις επιλογές για αλλαγές. Ήταν το συμβόλαιο αυτό μεταξύ της κυβέρνησής μας και των πολωνών πολιτών. Η δέσμευσή μας. Και από τη στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα, θέλησαμε να ελοπίσουμε αυτές τις αλλαγές, αυτές τις υποσχέσεις που είχαμε δώσει στους Πολωνούς, αυτές τις αλλαγές που επιθυμεί ο Πολωνός πολίτης για ριζική αλλαγή στο κράτος. Και το πράττουμε σεβόμενοι το Σύνταγμα, σεβόμενοι το νόμο και εν τέλει σεβόμενοι τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Και το επαναλαμβάνω. Είμαστε κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε, ήμασταν και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέρος αυτής της Ενωμένης Ευρώπης που προσφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους αυτό είναι το όραμά μας για την Ευρώπη. Θέλουμε μια Ευρώπη που σέβεται όλους τους Ευρωπαίους. Μια Ευρώπη που θα μεριμνά για τις εξελίξεις ολόκληρης της Ευρώπης. Και θέλουμε να είμαστε ενεργό μέλος μιας τέτοιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επί εκατοντοετίες έχει σέβεται η Πολωνία το κράτος δικαίου. είχε το πρώτο σύνταγμα της Ευρώπης με αξίες απαράβατες. Ένα σύνταγμα ιερό. Δεν παραβιάζουμε τη συνταγματική τάξη στη χώρα μου. Και θέλω να σας πω ότι χαίρομαι για την ευκαιρία που έχω σήμερα να σας παρουσιάσω την κατάσταση στην Πολωνία. Ωστόσο, οφείλω να επισημάνω πως δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να αφιερωθεί τόσος χρόνος και ενέργεια στα όσα συμβαίνουν στην Πολωνία πολλά άλλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα πρέπει ακόμα να επιληθούν, προβλήματα που αφορούν όλη την Ευρώπη ή άλλα κράτη της Ευρώπης. Εν πάση περιπτώσει όμως ας συζητήσουμε αυτά τα θέματα και επιτρέψτε μου να σας μιλήσω για τη χώρα μου για να σας εξηγήσω ό,τι χρήζει εξηγήσεως. Είμαι πεπισμένη, βαθύτατα πεπισμένη, ότι εάν και οι δύο πλευρές δείξουν ε, καλή διάθεση Βγαίνοντα από την αίθουσα αυτή, θα είμαστε πεπισμένοι πω η Πολωνία είναι χώρα ισχυρή που αναπτύσσεται ταχύτατα με τρόπο δυναμικό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι είναι μια χώρα για την οποία μπορούμε να είμαστε όλοι περήφανοι. Κυρίε και κύριοι, Για τι παρατηρήσει τώρα συγκεκριμένα για το Σταγματικό Δικαστήριο η πρώτη, για τα μέσα μαζική ενημέρωση η δεύτερη. Το Συνταγματικό Δικαστήριο, κυρίε και κύριοι, λειτουργεί άψογα στην Πολωνία είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Σήμερα μόλις, πριν από μερικές ώρες μάλιστα, το δικαστήριο αυτό εξέδωσε απόφαση, άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Οι αλλαγές που εισήχθησαν σε σχέση με τη λειτουργία του σταγματικού δικαστηρίου είναι σύμφωνες με το με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές δεν διαφέρουν δε σε τίποτα με αντίστοιχες διατάξεις άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Το νόμο για το σταγματικό δικαστήριο χρειάστηκε να τον τροποποιήσουμε για τον Ιούνιο του 2015 Ο προηγούμενος κυβερνητικό σχηματισμός είχε υιοθετήσει νόμο για το συνταγματικό δικαστήριο που είχε κριθεί αντισυνταγματικός από το ίδιο αυτό συνταγματικό δικαστήριο. Και άρα το ίδιο το συνταγματικό δικαστήριο είχε αμφισβητήσει τη συνταγματικότητα του νόμου αυτού που όπως είπα είχε υιοθετήσει η προηγούμενη κυβέρνηση, ο προηγούμενος κυβερνητικός συνασπισμός. Το ίδιο λοιπόν το συνταγματικό δικαστήριο είχε ζητήσει να διορθωθεί το σφάλμα. Οι δικαστές εκλήθησαν να λάβουν θέση αμέσως μετά τις εκλογές και εμείς προχωρήσαμε στην διόρθωση. 14 από 15 δικαστές έπρεπε να είχαν διοριστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η Επιτροπή της Βενετίας, στη γνωμοδότηση της οποίας στηρίζομαι εγώ το 1997, ορίζει πως το σύστημα επιλογής δικαστών στο Ανώτατο Σταγματικό Δικαστήριο θα πρέπει να στοχεύει σε καλύτερη δημοκρατική αντιπροσωπευτικότητα για το όργανο αυτό και ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να διορίζει δικαστές με βάση τις πολιτικές της επιλογές στο σύνολό τους. Αυτό το κανόνα θέλησαμε να εφαρμόσουμε. Ο νεοεκλεγής πρόεδρος μάλιστα είχε ζητήσει αλλαγή προς την κατεύθυνση αυτή και δεν δέχθηκε να ορκίσει δικαστές που είχαν με τον απατηλό αυτό τρόπο διοριστεί. Το Κοινοβούλιο λοιπόν υιοθέτησε την νομοθεσία προκειμένου να τροποποιηθεί η αντιδημοκρατική εκείνη ε, νομοθεσία που ε, όριζε τον τρόπο επιλογής και διορισμού των ε, δικαστών στο σταγματικό δικαστήριο, το οποίο είχε παραιτηθεί από την εξέταση επί της ουσίας των αποφάσεων αυτών. Έχουμε τώρα λοιπόν 15 δικαστές, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, στο Σταγματικό Δικαστήριο, που εκλέγονται, εκλέγονταν πάντα από την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Από αυτούς οι πέντε μόνο διορίστηκαν από την τρέχουσα κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Το κόμμα μας δεν θέλησε ποτέ ε, να ελέγξει το συνταγματικό δικαστήριο. Δεν επιδιώξαμε καν την πλειοψηφία των μελών του συνταγματικού δικαστηρίου να αντιστρέψουμε, να ανατρέψουμε. Θελήσαμε μόνο μια δημοκρατική λειτουργία. Οκτώ από τους 15 λοιπόν είναι διορισμένοι δικαστές, διορισμένοι από την τωρινή αντιπολίτευση. Και αυτή νομίζω είναι μια θετική διάκριση σε σχέση με την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς σεβόμαστε το δικαίωμα στο διάλογο. Και θέλουμε να συζητούμε και να παίρνουμε αποφάσεις από κοινού. Όπου υπάρχουν ζητήματα σοβαρά και κρίσιμα για την Πολωνία και τους Πολωνούς. Για να μπορέσει να εκδώσει μια απόφαση δημοκρατική θα πρέπει να συνέλθει και να ε, αποφασίσει στην ολομέλειά του το δικαστήριο. Όπως άλλωστε συμβαίνει και σε άλλα ευρωπαϊκά δημοκρατικά κράτη, όπου εκδικάζουν τις σοβαρές υποθέσει σε ολομέλεια τα σταγματικά δικαστήρια. Εμείς εισαγάγαμε την ιδέα της ειδική πλειοψηφία ή ενισχυμένης πλειοψηφία για τις αποφάσεις της ολομέλειας. Η πλειοψηφία που ισχύει και για την Εθνοσυνέλευση, όταν ε, συνέρχεται για να εγκρίνει νέο σύνταγμα, των δύο τρίτων δηλαδή, ισχύει και για το σταματικό Δικαστήριο. Υπάρχουν κράτη της Ευρώπης όπου απαιτείται αντίστοιχη απόλυτη πλειοψηφία για συγκεκριμένες υποθέσεις σταγματικού ε, τύπου από τα σταματικά δικαστήρια. Θα τα γνωρίζετε ασφαλώς. Πιστεύουμε ότι αυτή η δική πλειοψηφία θα επιτρέψει μια πιο συνταγματική, δημοκρατική λειτουργία του σταματικού δικαστηρίου. Πολλά άλλα επισημαίνονται σε σχέση με τις αποφάσεις του τελευταίου Δεκεμβρίου και πολλές παρεξηγήσεις υπάρχουν. Έχει δημιουργηθεί μια πολεμική που δεν είναι νομικής φύσεως αλλά πολιτικής. Το συνταγματικό δικαστήριο είναι ένα Δικαστήριο Δικαίου. Αποφασίζει κατά πόσο ένας νόμος για τον οποίο έχει προσφύγει κάποιος στο δικαστήριο θα διατηρηθεί και κατά πόσο κρίνεται συνταγματικός ή όχι. Οι νόμοι που το συνταγματικό δικαστήριο θεώρησε ότι δεν πρέπει να ισχύουν αποκλείστηκαν από το νομικό μας σύστημα. Αυτή είναι η μόνη νομική επίπτωση των αποφάσεων του συνταγματικού αυτού δικαστηρίου. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο για να κυρωθούν. Θέλω όμω επίση να υπογραμμίσω ότι σήμερα το δικαστήριο παίρνει και μια πολιτική διάσταση και δεν αποφασίζει μόνο επί της ουσίας. Αυτό είναι ένα δίλημα το οποίο πρέπει να λυθεί βάσει πολιτικού συμβιβασμού στην Πολωνία. Είναι εσωτερικό θέμα της Πολωνίας αυτό και πιστεύω ότι πρέπει να μας αφήσετε το πρόβλημα αυτό να το λύσουμε από μόνοι μας. Εγώ είμαι έτοιμη να το κάνω, είμαι έτοιμη να συζητήσω με την αντιπολίτευση και ελπίζω ότι οι λύσεις που θα προτείνουμε τελικά θα εγκριθούν από την αντιπολίτευση επίσης. Κυρίε και κύριοι, τώρα θέλω να αναφερθώ λίγο στι αλλαγέ στα δημόσια μέσα ενημέρωση, στα κρατικά μέσα ενημέρωση. Οι αλλαγέ αυτέ δεν πλήττουν καθόλου τι ευρωπαϊκέ προδιαγραφέ. Οι αλλαγές αυτές είναι προσπάθεια αποκατάστασης του αμερόληπτου χαρακτήρα των κρατικών μέσων ενημέρωσης στην Πολωνία. Μέχρι σήμερα, πολλοί λέγαν ότι δεν εξασφαλίζεται η ουδετερότητα, η αμεροληψία των μέσων ενημέρωσης. Χρειάζονταν λοιπόν αλλαγές για περισσότερο πλουραλισμό και για μεγαλύτερη ουδετερότητα είναι ο μόνος ο στόχος των αλλαγών που επιφέραμε. Πριν από τρεις εβδομάδες η πολωνική κυβέρνηση υιοθέτησε λοιπόν νόμο που τροποποιεί την νομοθεσία όσον αφορά τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Το Σώμα των Δημοσιογράφων της Πολωνίας ζήτησε την τροποποίηση αυτή και στο πρώτο στάδιο της μεταρρύθμισης εμείς διακανονίσαμε το θέμα που είχε να κάνει με τη διακυβέρνηση των κρατικών ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών σταθμών. Για να υπάρχει και κατάλληλη χρηματοδότηση. Χρειάστηκε λοιπόν να κατανείμουμε τις αρμοδιότητες ανάμεσα σε αυτούς που ορίζουν τα διευθυντικά στελέχη και τα συμβούλια επιτήρησης και ε, των άλλων που είναι στα όργανα που ρυθμίζουν άλλα πράγματα. Η Επιτροπή της Βενετίας του 2010 αναφέρει την υιοθέτηση τέτοιων μέτρων κατανομής αρμοδιοτήτων. Εδώ λοιπόν δεν έχουμε να κάνουμε με παραβιάσεις του συντάγματος, ούτε με θέματα παραβίασης των ελέγχων κλπ. Σήμερα η κυβέρνηση είναι στο δεύτερο στάδιο μεταρρύθμισης των κρατικών μέσων ενημέρωσης, προκειμένου τα μέσα αυτά να έχουν την κατάλληλη και σταθερή χρηματοδότηση. Αυτό που μας εμπνέει εδώ είναι οι λύσεις που ισχύουν σε πάρα πολλές χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, η κυβέρνηση της πολωνικής δημοκρατίας είναι ανοιχτή σε διάλογο και σε συζήτηση. Εμείς θέλουμε σε συνεργασία με όλες τις πλευρές στην Πολωνία αλλά και αλλού να έχουμε επικοδομητικό διάλογο. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τα πολιτικά κόμματα της αντιπολίτευσης και με όσους σήμερα στηρίζουν την δράση της πολωνικής κυβέρνησης. Θέλουμε να επιφέρουμε θετικές αλλαγές στην Πολωνία. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν στη συζήτηση, ανοιχτοί στο διάλογο και θέλουμε μαζί από κοινού να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα. Αυτό που είναι πάνω απ' όλα σημαντικό είναι ότι θέλουμε να νιώθουμε τη στήριξη των άλλων χωρών. Θέλουμε να έχουμε την εντύπωση ότι η Πολωνία ως ελεύθερη και κυρίαρχη χώρα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να βασίζεται στη στήριξη των άλλων χωρών. Και όταν πρόκειται για αποφάσεις που αφορούν το εσωτερικό της χώρας, θα έχουμε την εγγύηση ότι τηρείται η εθνική μας κυριαρχία και ότι τη σέβεστε. Είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε σε ό,τι ερωτήσεις έχετε και να σας δώσουμε ό,τι επιπλέον πληροφορίες θέλετε. Και εγώ και τα μέλη της πολωνικής κυβέρνησης. Η Πολωνία είναι μια όμορφη χώρα. Η Πολωνία είναι ένας περήφανος λαός. Εμείς θέλουμε να είμαστε πρωταθλητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το όνειρό μας. Αυτό είναι το όνειρο των Πολωνών. Περιμέναμε πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ για να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε και εμεί να υποφεληθούμε και να χαρούμε από τη δημοκρατία και από τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σήμερα δεν μπορούμε να παραιτηθούμε από τις αρχές αυτές τι τόσο σημαντικές για μας. Δεν υπάρχει τίμημα για όλα αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας λοιπόν και είμαι βαθιά πεπισμένη ότι μετά από τις εξηγήσεις αυτές που σας έδωσα θα σκεφτείτε τα πράγματα βάσει αυτών των νέων πληροφοριών και θα καταλήξετε στα συμπεράσματά σας. Είμαι πεπισμένη ότι μέσω του διαλόγου θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε ένα καλό μέλλον για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρωθυπουργέ εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριο Κονσάλε Πόνς. Κύριε Πρωθυπουργέ, ο πρόεδρος της ομάδας μου, ο κύριος Βέμπερ, είναι Γερμανός. Έτσι, με κάθε σεβασμό, μου ανέθεσε εμένα, μου έδωσε τη θέση του, δηλαδή για να μην μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει σαν άλλο την εθνικότητα, την προέλευση. Κύριε Πρωθυπουργέ, η δεύτερη μεγαλύτερη αντιπροσωπεία στην ομάδα μας είναι η Πολωνία, αλλά δεν είναι οι Πολωνοί που θα σας απαντήσουν, γιατί κανένας δεν θέλει να χρησιμοποιηθεί σαν άλοθη η εθνικότητα. Κύριε Πρωθυπουργέ, δεν είναι λογικό στην Ευρώπη να παίρνουμε τα μέτρα μας προκειμένου τα λόγια να μην χρησιμοποιούνται σαν όπλα. Σας μιλάει λοιπόν ένας Ισπανός, ένας Ισπανός από το ΕΛΚΑ. Στη θέση μου όμως θα μπορούσε να ήταν οποιοδήποτε από την ομάδα μου, γιατί όλοι πιστεύουμε τα ίδια. Η Ευρώπη πριν από οτιδήποτε άλλο είναι ένα σύνολο δημοκρατικών αξιών. Και στη συνέχεια είναι μια αγορά. Επαναλαμβάνω, πρώτα είναι μια κοινότητα αξιών και μόνο μετά είναι μια αγορά. Γι' αυτό εκ μέρου όλων θέλω ναι, έχω τη βεβαιότητα ότι και εσείς συμφωνείτε με αυτό, ότι η Ευρώπη δηλαδή δεν είναι οι Βρυξέλλες, δεν είναι το Βερολίνο, δεν είναι το Παρίσι. Ευρώπη είμαστε 500 εκατομμύρια άνθρωποι που θέλουμε να συνεπάρξουμε. Οι Πολωνοί αγωνίστηκαν κατά όλων των δικτατοριών και τις νίκησαν, κατά του ρατσισμού επίσης. Εμείς είμαστε με την Πολωνία στη συνέχεια κατά του κομμουνισμού και οι Ευρωπαίοι σταθήκαμε στο πλευρό των Πολωνών. Σήμερα όλοι οι Ευρωπαίοι αγωνιζόμαστε κατά της τρομοκρατίας. Όμως ο αυταρχισμός δεν έρχεται πάντα απ' έξω. Ο αυταρχισμός δεν γνωρίζει ούτε εποχές, ούτε τόπους, το θέμα είναι να στηρίξουμε τις αξίες μας και τις ελευθερίες μας. Οι Πολωνοί γνωρίζουν δυστυχώς πολύ καλά, όπως και οι Ισπανοί, όπως και οι Πορτογάλοι, όπως και οι Ιταλοί, όπως οι Γερμανοί, όπως οι Ρουμάνοι, οι Σλοβαίνοι, οι Γάλλοι, οι Έλληνες. Γνωρίζουν ότι ο χειρότερος αυταρχισμός έρχεται απ' έξω και από μέσα όμως είναι μια βασική αρχή αυτή στην οποία πρέπει να πιστέψουμε ο αυταρχισμός οδηγεί στην κατάργηση της δημοκρατίας. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι Πολωνία, είναι ο αυταρχισμός, ο οποίος δημιουργείται όπου δημιουργείται. Τα σφάλματα του παρελθόντος πρέπει να τα αποφύγουμε. Ακόμα και οι μεγαλύτερες φρικαλαιότητες πρέπει να αντιμετωπιστούν, να μην τις ξαναζήσουμε ποτέ. Όλοι μαζί, ενωμένοι. Η Ευρώπη βασίζεται στη συμφιλίωση, όχι στην εκδίκηση. Εμείς θέλουμε τις ανθρώπινες αξίες. Η Ευρώπη βασίστηκε στο ρωμαϊκό δίκαιο και στην ε, χριστιανική αντίληψη. Αυτό συζητάμε σήμερα. Θέλουμε να διευκρινίσουμε κατά πόσο υπάρχει δυνατότητα κάποια από αυτές τις αξίες να διακινδυνεύει ή όχι. Σήμερα κανένας δεν έρχεται ούτε να κατηγορήσει, ούτε να καταγγείλει, ούτε να καταδικάσει. Συζητάμε για δράσεις και Κυρία Πρωθυπουργέ, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκαθαριστούν οι παρεξηγήσεις, αν χρειάζεται και αν υπάρχουν παρεξηγήσεις. Κανείς δεν θέλει να καταδικάσει προληπτικά την πολωνική κυβέρνηση και λιγότερο από οποιοδήποτε άλλους το ΕΛΚ. Οι Πολωνοί του ΕΛΚ ποτέ δεν θα δοκίμαζαν κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν αναμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα του διαλέγου αυτού και ζητάω από τους επιτρόπους και αυτοί πολύ προσεκτικά να παρακολουθήσουν την κατάσταση. Όταν πρόκειται για εσωτερικά ζητήματα, κυρία Πρωθυπουργέ, εννοείται ότι έχετε κάθε νομιμότητα και είναι απόλυτα θεμητό να υλοποιήσετε το κυβερνητικό σας πρόγραμμα όπως πιστεύετε εσείς. Θα σας κρίνουν οι Πολωνοί ψηφοφόροι σας. Αυτό όμως που μας επηρεάζει όλους είναι το κράτος δικαίου δεν πρέπει, αγαπητοί φίλοι, να ξεγελιόμαστε. Οι, ως καλή εταίροι πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια και πρέπει να λέμε ένας στον άλλον την αλήθεια. Όπως είπαμε την αλήθεια στην ελληνική κυβέρνηση, όπως λέμε την αλήθεια στους Βρετανούς, στη Βρετανική κυβέρνηση. Έτσι και σήμερα εδώ, εσείς και εμείς θα μιλήσουμε και θα πούμε την αλήθεια. Θα πούμε τα πράγματα όπως έχουν. Κυρία Πρωθυπουργέ, δεν πρόκειται για τον νόμο, πρόκειται για τις αξίες. Εσείς λοιπόν, όπως οποιαδήποτε νόμιμη κυβέρνηση, μπορείτε να αλλάξετε τον νόμο. Αλλά ούτε εσείς ούτε καμία νόμιμη κυβέρνηση δεν μπορεί να αλλάξει τις αξίες. Ποτέ, κυρία Πρωθυπουργέ. Εκ μέλους της ε, ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, ο κύριος Πιτέλα. Οι οι σοσιαλιστές και δημοκράτες αναμφίβολα βρίσκονται στο πλευρό των χιλιάδων Πολωνών που κατέβηκαν στους δρόμους αυτές τις εβδομάδες για το κράτος δικαίου και την δημοκρατία. Κυρία Πρωθυπουργέ, εδώ βρίσκομαι. Κυρία Πρωθυπουργέ, εκτιμώ με τον, ε, το ύφος της παρέμβασής σας. Και δεν θέλουμε να περάσουμε από δίκη την Πολωνία. Ούτε να αντιστρέψουμε την δημοκρατική πορεία και κατεύθυνση της χώρας σας. Εσείς έχετε αναλάβει πλήρη καθήκοντα, με πλήρη αυτονομία, να κυβερνήσετε τη χώρα σας με τις επιλογές που εσείς προκρίνετε. Όμως με πλήρη σεβασμό των αρχών και των αξιών του ευρωπαϊκού δικαίου. Η Πολωνία είναι ένας από τους πυλώνες της Ένωσης και ιστορικός και λόγω του ε, παρελθόντος της και λόγω του αγώνα της κατά των απολυταρχικών καθεστώτων. Στον 20ο αιώνα ο πολωνικός λαός είναι παράδειγμα για όλους μας. Τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει, η κυβέρνησή σα, ε, κυρία Πρωθυπουργέ, δυστυχώ αρνούνται και αντιφάσκουν με αυτή την ιστορία ελευθερία. Έναν εξάρτητο συνταγματικό δικαστήριο και μέσα επικοινωνία ελεύθερα είναι προποθέσει για το κράτο δικαίου. Έτσι θεωρήσαμε επίκαιρη και δίκαιη την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την ευχαριστούμε όλους ιδιαίτερως. Ευχαριστούμε τον Αντιπρόεδρο Τίμερμανς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προξενιό, ούτε γάμος ε, συμφέροντος, ούτε από τράγος. Είναι μια ένωση αξιών, ελευθεριών και δημοκρατίας. Ε, η Ευρώπη χρειάζεται μια Πολωνία ελεύθερη και ισχυρή. Ε, στοχαστείτε το, κυρία Πρωθυπουργέ. Σκεφτείτε τι μέτρα εγκρίνατε και δεχτείτε τον διάλογο και την ε, αντιπαράθεση απόψεων, όπως είπε προηγουμένως και ο πρόεδρος Τίμερμανς. Η Πολωνία είναι μια χώρα μεγάλη και εμείς δεν θα την αγκαταλείψουμε μην την κατευθύνετε σε μία οδό που δεν είναι αντάξια της ιστορίας και της παράδοσής της. Ευχαριστούμε. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Καμάλη. Ευχαριστώ πολύ. Καθώς βρισκόμαστε εδώ σήμερα το απόγευμα, διαισθάνομαι ότι οι ευρωβουλευτές προσπαθούν ε, να δουν, ε, να βρουν σχόλια καθησυχαστικά για την πολιτική κυβέρνηση. Αλλά α πάρουμε λίγο απόσταση και α σκεφτούμε ότι η Επιτροπή τη Βενετία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν να συνεργαστούν με την πολωνική κυβέρνηση και να διασκεδάσουν εκείνη τι ανησυχίε μα. Έχω μιλήσει με την Πρωθυπουργό και πολλού υπουργού νωρίτερα σήμερα και είναι σαφέ ότι δεν έχουν καμία ε, πρόθεση να υπονομεύσουν την πολυφωνία και το κράτο δικαίου. Γιατί όταν η τελευταία κυβέρνηση αποφάσισε προτού αφήσει τα καθήκοντά τη να διορίζει του δικού τη δικαστέ, δεν ξεκίνησε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, έρευνα για το θέμα αυτό και οι ευρωβουλευτέ δεν διαμαρτυρήθηκαν. Γιατί μόλι η νέα κυβέρνηση διόρισε πέντε από του 15 δικαστέ του Συνταγματικού Δικαστηρίου έχει γίνει αυτό ο άλλο. Θα πρέπει να έχουμε επικοδομητικές ε, συνομιλίες και να εκτιμήσουμε την ε, στάση της ε, πολωνικής κυβέρνησης. Θα πρέπει να ζητήσουμε την άποψη της κυβέρνησης και να χαρούμε για την διάκριση που έκανε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταξύ ρυθμιστού και ραδιοτηλόρασης. Θα πρέπει αυτό να γίνει και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε στα τηλεοπτακουστικά, και όταν ασχολήθηκα με την οδηγία που είχε ακριβώς αυτό το θέμα, πραγματικά σοκαρίστηκα από τον αριθμό ευρωβουλευτών βουλευτών από τα νέα κράτη-μέλη που ήταν και μέλη Συμβουλίου τηλεοπτικού της χώρας τους. Αυτό αποτελεί σύγκρουση συμφερόντων και στην αίθουσα εδώ υπάρχουν πρώην εθνικοί πολιτικοί που ήταν εκδότες εφημερίδων ή δούλευαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς και ήταν όχι συντάκτες και κάποιοι από, αυτές, από αυτούς αποφάσιζαν ποιος θα απολυθεί και ποιος όχι. Εάν λοιπόν θέλουμε σήμερα να αμφισβητήσουμε την νόημα εκλεγμένη πολωνική κυβέρνηση είναι σαν να διεκδικητούμε τους ανθρώπους που την ψήφισαν, τους ίδιους τους Μην εκπλαγείτε λοιπόν εάν οι Πολωνοί τελικά εκλέξουν περισσότερους ευρωσκεπτικιστές όπως την Ιταλία, τη Γαλλία και την Ουγγαρία. Εδώ λοιπόν θα καλέσω όλους να είναι προσεκτικοί στις εκφράσεις τους. Όταν ε, έγιναν σχόλια εδώ στο Κοινοβούλιο από τους ε, Γερμα... Όταν ο, ο κ. Μπερλουσκόνη λοιπόν έκανε σχόλια εδώ προς τον κ. Σούλτ για το παρελθόν ε, της Γερμανίας, εδώ πέρα ξέσπασε διαμαρτυρία Οπότε πρέπει να σκεφτούμε πώ εδώ μπορεί να προσβάλλουμε τον πολωνικό λαό, οι οποίοι έπρεπε να αντιμετωπίσουν τις, το ρωσικό υπερελισμό, τον κομμουνισμό, και ε, να ε, ξεπεράσουν ε, τις απειλές και πιέσεις που έχουν δεχτεί ως τώρα. Ας δούμε τις πραγματικές κρίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ. Την μετανάστευση, την κρίση του ευρώ και τη χαμηλή ανάπτυξη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταλήξει σε πορίσματα βάσει δίκαιων αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων και λαμβάνοντα υπόψη την ιστορική οδύνη του πολωνικού λαού που τόσες φορές έχει πέσει θύμα άλλων δυναστών. Να έχουμε λοιπόν υπόψη όλα αυτά τα στοιχεία και ε, την πολιτική κυβέρνηση να την αφήσουμε να συνεργαστεί μαζί μας γνωρίζοντας ότι και εμείς πρέπει να δείξουμε συνεργασία και πνεύμα συνεργασίας. Να σεβαστούμε την ελευθερία, την ελευθερία έκφρασης και τη δημοκρατία για την οποία ο πολωνικός λαός αγωνίστηκε τόσο σκληρά. εκ μέρους των φιλελευθέρων ο πρόεδρος κ. Φερχόφστατ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρωθυπουργέ, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και πάνω απ' όλα για τον τόνο που ε, χρησιμοποιήσατε. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω και εγώ το δικό σας παράδειγμα. προς τον τόνο, πράγμα που βέβαια δεν συνηθίζω, δεν είναι εύκολο δηλαδή για μένα. Εσείς όμως και το κόμμα σας κερδίσατε εκλογέ. Εσείς και το κόμμα σας λάβατε ισχυρή εντολή να ηγηθείτε της χώρας. Το σεβόμαστε αυτό, όπως οφείλουμε να το σεβαστούμε ως ε, φιλελεύθερος μπορεί να μην με συμφωνώ με όλες τις πολιτικές σας. Αλλά η δημοκρατία αυτό προβλέπει. Και με βάση την πλειοψηφία που κερδίσατε έχετε το δικαίωμα να διαμορφώσετε το μέσο ε, μαζικής ενημέρωσης, τη δημόσια διοίκηση. Να σας πω, και εγώ ε, διατέλεσα πρωθυπουργός και έκανα και εγώ τέτοια αντίστοιχα. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, αυτό που μας ανησυχεί, αυτό που ανησυχεί όλους τους να συναδέλφους εδώ, είναι, και αυτό που δεν κάνει ποτέ ένας δημοκράτης, είναι να αξιοποιεί ή να καταχράται αυτή της πλειοψηφία για να ανατρέψει ισορροπία στη χώρα. Αυτό είναι που δεν συμβαίνει ποτέ. Γιατί, Γιατί αυτή είναι η καρδιά της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Το σύστημα αυτό των ισορροπιών δυνάμεων που επιτρέπει να εισάγονται νόμοι ακόμη και όταν αυτοί είναι σε αντίθεση με το Σύνταγμα της Πολωνίας. Η πλειοψηφία σας, νομίζω ανήμερα των Χριστουγέννων, έσπευσε να περάσει αυτή την νομοθεσία για το σταγματικό δικαστήριο που ουσιαστικά το αδρανοποιεί. Και σας επισημαίνω ότι δεν το είχατε περιλάβει στο μανιφέστο σας το προεκλογικό. Θα είμαι δε πολύ συγκεκριμένος. Το ζήτημα δεν είναι η σύνθεση, οι διορισμοί, κυρία Καλά, Καμάλ. Δεν είναι ο αριθμός, δεν είναι η πλειοψηφία των δύο τρίτων ε, που επιβάλλατε, ούτε καν η χρονολογική σειρά του πινακίου που έχετε εισαγάγει ως κανόνα. Το είπατε εσείς άλλωστε. Κάποιοι κάποια κράτη-μέλη έχουν τέτοιου κανόνες. Ναι, αλλά δεν έχουν τον συνδυασμό αυτών των κανόνων. Ο συνδυασμός των τεσσάρων αυτών στοιχείων ταυτόχρονα οδηγεί σε παράλυση το δικαστήριο, το καθιστά ανίκανον επιτελέσει το έργο του. Και κύριε Καμάλ, ναι, μπορεί η πολωνική κυβέρνηση να έχει διορθώσει λάθος σφάλματα τη προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά δεν διορθώνεται λάθη στην ουσία παρα, οδηγείται σε παράλυση το Σταγματικό Δικαστήριο. Από τον τόνο δε της ομιλίας σας εγώ ε, διαβάζω, από τη φωνή σας ακόμα, πως βλέπετε πρόβλημα. Και γι' αυτό δεχθήκατε τις συμβουλές του κυρίου τις καλές συμβουλές, να ε, ζητήσετε γνωμοδότηση από την Επιτροπή της, της Βενετίας. Αλλά θα ήταν μεγάλο σφάλμα να σπρώξουμε την Πολωνία προς Ανατολάς, προς άλλο σύστημα διακυβέρνησης. Ναι, ξέρω κύριε Καμάλ, ε, αναφορά στον Πούτιν. Ξέρω ότι του κυρίου Κασίνσκι δεν του αρέσει ούτε ο Πούτιν ούτε η Ρωσία. Ούτε και εμένα βέβαια γιατί είμαι και στη μαύρη λίστα. Αλλά με τις πολιτικές αυτές, είπα εγώ, ο κύριος Κασίνσκι βοηθάει τον κύριο Πούτιν. Γιατί η δυσάρεστη αλήθεια είναι ότι ο κύριος Πούτιν δεν θέλει την Ευρωπαϊκή Ενότητα. Τουναντίον έχει μονομανία να καταστρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα τακτενόμενα στην Πολωνία μπορεί να τον βοηθήσουν σε αυτό το στόχο του. Μην ξεχνάτε κυρία Πρωθυπουργέ, η ιστορία έχει αποδείξει πως η ενότητα και η ισχύ της Πολωνίας βαίνουν χέρι με χέρι με την ευρωπαϊκή ενότητα και με την ευρωπαϊκή ισχύ, με την ισχύ της Ευρώπης διαχρονικά δεν έχω καμιά αμφιβολία, έχω κάθε εμπιστοσύνη στον, Ευρω... στον πολωνικό λαό, στον πολωνό πολίτη. Θυμάμαι πώς αγωνίστηκε με τη Σολινταρνόσκ κατά της καταστολής, για τις ελευθερίες, για τη δημοκρατία, για την ελευθερία της θρησκευτική πίστης, για το κράτος δικαίου. Για όλα αυτά αγωνίστηκε ο πολωνικός λαός και είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται ποτέ να παρετηθεί από τη δημοκρατία του. Και γι' αυτό η έκκλησή μου προς εσάς, κυρία Πρωθυπουργέ, η έκκλησή μου προς εσάς, δεν θέλω να σας καλέσω, όχι τόσο να ακούσετε εμένα ή εμάς εδώ, ακούστε αφού την πλειοψηφία των πολιτών σας, αυτών που θέλουν και στο μέλλον να μείνει αυτή η χώρα στην παγκόσμια κοινότητα των δημοκρατιών. Ευχαριστώ πολύ. Για την Ανωτική Αριστερά η πρόεδρος της κυρία Τσίμερ. Αξιότιμη κυρία Πρωθυπουργέ, κυρία Σίτλο, ευχαριστώ πολύ που ήρθατε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα για να ε, συζητήσετε για το κρίσιμο αυτό θέμα. Είστε βεβαίως αρχηγός κυβερνήσεως και έχετε δικαίωμα και υποχρέωση να εκτελείται καθήκοντα, καθήκοντα σταγματικής τάξης. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ελευθερία, η δημοκρατία, κράτος δικαίου, η ε, διαφύλαξη των ανθρωπινών δικαιωμάτων υπόθηκε εδώ, είναι συγκαταλεγόντα μεταξύ των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό απαιτεί ανεξάρτητα δικαστήρια και ανεξάρτητα μέσα ε, ενημέρωσης ταυτόχρονα. Εξού και η ερώτηση που σας απευθύνεται και χαίρομαι που είπατε ότι θα δεχθείτε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας και σχετική συζήτηση, άρα θα τα ξαναπούμε. Και επίσης χαιρόμαστε για το ότι έχει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία επαλήθευσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. διαδικασία επαλήθευσης, η οποία πιστεύω εφαρμόζεται για πρώτη φορά, δεν υπήρχε στο παρελθόν με αυτή τη μορφή, διαδικασία επαλήθευσης η οποία θα έπρεπε Καταρχήν και κάθε φορά όπου ε, γεννώνται ζητήματα, αφιβολίες ε, ανησυχίες σε σχέση με ένα κράτος μέλος και ανεξαρτήτως του κράτους μέλους και της πολιτικής πλειοψηφίας στο κράτος αυτό, θα έπρεπε να γίνεται αυτή η επαλήθευση με ένα διαρθρωτικό ουσιαστικό διάλογο. Το ζήτημα δεν είναι ε, η δημοκρατική νομοποίηση της πολωνικής κυβέρνησης, αλλά η δημοκρατικότητα των δράσεων και των πράξεων σας. Και σε αυτό θέλουμε να περιορίσουμε τη συζήτηση. Τα προβλήματα, και θέλω επίσης να επισημάνω ότι δεν ε, είναι ουρανοκατέβατα, νεοφιλελεύθερες, ακόμη και ακραίες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που κατέστησαν απαραίτητες για την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εξασφάλισαν με την ε, χρόνο ευημερία για όλους και τα ανθρώπινα δικαιώματα παραγνωρίστηκαν πολλές φορές. Πολύ είναι αυτοί στην Πολωνία αλλά και σε άλλα ανατολικοευρωπαϊκά κράτη οι οποίοι δεν μπόρεσαν να ε, συζητήσουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της δημοκρατίας, της ε, δικαιοσύνης της ελευθερίας. Δέχθηκαν την Ευρωπαϊκή Ένωση σαν ένα, υπο, σαν έναν οργανισμό ε, υπεύθυνο και για τα κοινωνικά προβλήματα στα οποία οδηγήθηκαν. Και τώρα βεβαίως λέτε ότι διαφοροποιήστε σε σχέση με τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Υπήρχε η κυβέρνηση πριν, φιλελεύθερη, η οποία επί παραδείγματι δεν συζήτησε, δεν έθεσε ως ζήτημα συζήτησης την καταπολέμηση της φτώχειας. Και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά στην Ευρώπη. Τα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα πρέπει να ισχύουν για τους πάντες στην Ευρώπη. Θέλετε η Πολωνία να είναι πρωταθλήτρια μες στην Ευρώπη. Μακάρι. Εγώ δεν θέλω να έχει ηγετικό ρόλο η Γερμανία. Εγώ θέλω όλοι να συνεργάζονται. Τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης, Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης που προσχώρησαν το 2004 και έχουν πολύ έδαφος να καλύψουν, αλλά έχουν και πολλά να προσφέρουν ακόμη, να προχωρήσουν ακόμη περισσότερο. Έχουν γίνει μεγάλα σφάλματα στην ε, διαδικασία αυτή της προσχώρησης και της Ενωπής Ευρώπης. Εάν θέλετε να είστε προς πρωταθλήτρια στην Ευρώπη, διαρωτηθείτε τι στάση θα έχετε σε σχέση με τη μετανάστευση. Δεν μπορεί η Πολωνία να λέει εφέτος μόνο 400 Παρακαλώ, ξανασκεφτείτε το. Πρώτο ερώτημα. Και δεύτερο, η Πολωνία έχει ε, αυτοεξαιρεθεί με το opt-out από τον χάρτη των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Δεν θα ήταν πολύ καλό μήνυμα να αναστέλατε αυτή την αυτοεξαίρεση και έτσι να επιτρέπατε στους Πολωνούς πολίτες να τύχουν της, ε, του σεβασμού και αυτού του χάρτη των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Ο πρόεδρος, η κυρία Χάρμς, εκ μέρους των Πρασίνων. Κυρία Πρωθυπουργέ, θα αντιληφθήκατε φαντάζομαι ότι η σημερινή συζήτηση περιστρέφεται περί της ε, ανησυχίες και τα τεκτενόμενα στην Πολωνία, το κράτος δικαίου στην Πολωνία, αλλά Φαντάζομαι θα έχετε διαγνώσει πίσω από τη συζήτηση αυτή τις ε, ανησυχίες μας για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για το ότι δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου, ότι δεν υπάρχει σεβασμός στο κράτος δικαίου. Υπόθηκε αυτό ήδη. Η εσωτερική αγορά, η νομοθεσία, οι εγγυήσει για τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Τίποτα δεν λειτουργεί σωστά στην Ευρώπη εάν δεν γίνεται σεβαστό το κράτος δικαίου και πολύ σωστά μας υπενθυμίσατε τη σημασία, το ρόλο του πολωνικού έθνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την διαμόρφωσή της, την τωρινή της μορφή. Ως ε, πολιτιολόγος για θέματα, ε, ως ε, πολιτικός Ευρωπαία θα ήθελα να επισημάνω τα λόγια σας. Είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε όμως. Ήταν σωστό η Πολωνία και τα άλλα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει αμφισβητηθεί αυτό. Εγώ έχω τελείως διαφορετική γνώμη και οι αγώνες των Πολωνών στο δικό μου τον εσωτερικό απολογισμό, εκείνο το μαγικό Αύγουστο του 1980, σηματοδότησε ένα σημείο καμπή δική μου τη ζωή, γιατί αγωνίστηκαν όχι μόνο για την ελευθερία και τη δημοκρατία, για την Πολωνία οι Πολωνοί το 1980, αλλά για τη δημοκρατία, τη σταθερότητα και την ασφάλεια σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το φίλμα στους Πολωνούς. Έχω λοιπόν κάθε εκτίμηση για αυτούς τους αγώνες, ωστόσο και γι' αυτόν ακόμα το λόγο, ακόμη περισσότερο, πολύ δύσκολα δέχομαι τα όσα βλέπω να εξελίσσονται στην Βαρσοβία από τότε που αναλάβατε εσείς την εξουσία. Από αυτά που ακούω όχι από κάποιους έμεσους, κάποιες έμεσες πηγές, αλλά από τους ίδιους τους πολίτες της ε, Πολωνίας, που δεν είναι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφέρω τον Ματέο Σκιώφσκι, ο οποίος ήρθε ειδικά σήμερα στο Στρασβούργο για να ε, προσωπήσει μια πολύ σημαντική και διαφορετική θέση. Κυρίες και κύριοι, ο Γκίφερ Χόφστατ επεσήμανε και περιέγραψε σωστά τα προβλήματα σε σχέση με το κράτο δικαίου. Δεν πρόκειται για αποφάσει που αφορούν πρόσωπα. Πρόκειται για την εντύπωση πω μια κυβερνητική πλειοψηφία επιβάλλει με διατάγματα, αποφάσεις. Μέσα σε μια νύχτα πήρατε αποφάσεις οι οποίες χρειάζονται πολύ τη συζήτηση κανονικά. Η δική μου πολιτική ομάδα θεωρεί ότι αυτός ο μηχανισμός κράτου δικαίου, κράτους δικαίου που είδαμε να αναπτύσσεται σε σχέση με την Ουγγαρία θα πρέπει να αξιοποιηθεί, αλλά πάνω απ' όλα θα πρέπει οι αποφάσεις να ληφθούν στο τέλος του διαλόγου όχι να γίνεται λόγος, όπως κάνουν ορισμένοι Γερμανοί συναδελφοί, για κυρώσεις από τώρα. Και επίσης, το ζήτημα μιας επιλεκτικής αντιμετώπισης. Εμείς ως ομάδα των Πρασίνων πάντα υποστηρίζαμε πως χρειάζονται εργαλεία για την επαλήθευση τη λειτουργία του κράτου δικαίου, των εγγυήσεων του κράτου δικαίου, γιατί αυτό είναι ο συνδετικό ιστό τη Ευρώπη. Αυτό όμω, το, το οποίο δεν δεχόμαστε είναι για αλλητικών συμφερόντων κάποιους να τους προστατεύουμε και να παραγνωρίζουμε για λόγους κομματικούς τα προβλήματα σε επίπεδο κράτους δικαίου. Η Επιτροπή της Κοπεχάγης πρέπει να μετατραπεί σε μια συμβουλευτική επιτροπή η οποία θα ε, δρά κατά της επιλεκτικής επίδειξης ορισμένων προβλημάτων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος και διακόπτη. Εκ του Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι. Είμαι ο πρώτος Πολωνός Ευρωβουλευτής που παίρνει το λόγο σε αυτή τη συζήτηση και θέλω να υπογραμμίσω ότι τα πολωνικά ζητήματα πρέπει να λύνονται στην Πολωνία από Πολωνούς. Λυπούμε λοιπόν που κάποιοι δεν μπορούν να δεχτούν τα αποτελέσματα των πολωνικών εκλογών. Η συζήτηση αυτή η σημερινή δεν έχει λόγο ύπαρξης. Όπως είπε και η Πρωθυπουργό στην παρέμβασή της, θα υπάρξουν πλεονεκτήματα τελικά από αυτή τη συζήτηση, γιατί θα αυξηθούν οι ευρωσκεπτικιστές στην Ευρώπη. Οι Ιταλοί, οι Γερμανοί και άλλοι γίνονται όλο και περισσότερο κατά τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί δεν ανταποκρίνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ρόλο της στο λόγο για τον οποίο δημιουργήθηκε και δεχόμαστε παρεμβάσεις από το εξωτερικό. Πριν από 200 χρόνια η Ρωσία, η Προσία και η Αυστρία ασχολήθηκαν με την τύχη της Πολωνίας, κάτι το οποίο οδήγησε στην εξαφάνιση της χώρας της Πολωνίας, δηλαδή για δεκαετίες. Πριν όμως από μερικά χρόνια τελικά καταφέραμε να βγούμε από το κομμουνιστικό σύστημα και πάλι θέλαν να παίξω να μας βοηθήσουν. Σήμερα είναι οι Ευρωπαίοι Επίτροποι που θέλουν να μας βοηθήσουν. Όχι, οι Πολωνοί είναι αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν με τα πολωνικά ζητήματα και κανένας άλλος. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Μαρούζικ, εκ μέρους της Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κύρια Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για αυτά που άκουσα από τον συνάδελφο. Με τον ίδιο τρόπο σκέφτομαι κι εγώ. Παίρνω το λόγο λοιπόν ως μέλος της πολιτικής μου ομάδας, αλλά και ως Πολωνός. Και εγώ ως Πολωνός δεν ανησυχώ καθόλου για την κριτική που ακούγεται απ' έξω για τη χώρα μου. Μάλιστα, αυτό θα μπορούσε και να σημαίνει ότι τα μέτρα που υιοθετεί η πολωνική κυβέρνηση συνάδουν με τα, με τα πολωνικά συμφέροντα. Με ικανοποιεί αυτό, ούτε και ανησυχώ για τις αρνητικές απόψεις που εκφράζονται εδώ στο ημικύκλιο, γιατί δεν επηρεάζουν καθόλου την πολωνική κατάσταση. Εμείς θέλουμε στην Πολωνία να λύσουμε τα προβλήματά μας. Αυτό όμως που βρίσκω προβληματικό είναι ότι η σημερινή συζήτηση λαμβάνει χώρα. Αυτό είναι το πρόβλημα της Ευρώπης. Αυτή η συζήτηση δεν έχει λόγο ύπαρξης. Δείχνει την ανάμειξη. Πώς απ' έξω θέλει η Ευρώπη να αναμειγνύεται στα εσωτερικά των χωρών μελών. Και αυτή είναι η κατάρα της Ευρώπης. Στη συζήτηση αυτή τελικά τίποτα δεν μπορούμε να πούμε για την πολιτική κατάσταση στην Πολωνία. Αυτό που δείχνει η συζήτηση αυτή είναι την πολιτική καταστροφή. Μέσα σε αυτή την πολιτική καταστροφή βρίσκεται η Ευρώπη σήμερα αποτελεί διέξοδο η συζήτηση αυτή για την Ευρώπη, γιατί η Ευρώπη θέλει να αποφύγει τα δικά της τα προβλήματα, τα προβλήματα τα δικά της που δεν είναι σε θέση να λύσει. Ως μέλος λοιπόν της πολιτικής ομάδας της Ευρώπης των Εθνών και της Ελευθερίας, σας λέω ότι το σχέδιο αυτό το ευρωπαϊκό είναι νεκρό. Προχωράει μόνο λόγω αδράνειας, τίποτα άλλο. Για να διορθωθεί η Ευρώπη θα έπρεπε να διασφαλίσει την προστασία μας και θα έπρεπε να βρει έναν άλλο τρόπο συνεργασίας κυρίαρχων εθνών μέσα στην Ευρώπη. Αυτό πρέπει να κάνουμε και αυτό οφείλουμε στους συμπολίτε μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Κόρβιν Μίκε. Μη γεγραμμένος. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ μισώ τη δημοκρατία. Εσείς όμως είσαστε δημοκράτης. Λοιπόν, οι Πολωνοί εξέλεξαν σύμφωνα με τον νόμο και απολύτως δημοκρατικά το κόμμα το οποίο βρίσκεται σήμερα στην κυβέρνηση δικαίου και δικαιοσύνης. Το κόμμα αυτό λοιπόν δικαίου και δικαιοσύνης χάρη της πλειοψηφίας που τον έδειξε στην κυβέρνηση, θα κάνει αυτό που πιστεύει ότι είναι σωστό. Αν πιστεύετε ότι είναι κακό αυτό το κόμμα, εντάξει, συμφωνώ μαζί σα. Αλλά και η προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ακόμα πιο κακή. Θυμηθείτε τη διαφθορά, θυμάτε, θυμηθείτε μάλλον τον τρόπο με τον οποίο καταπιέζονταν η ελεύθερη έκφραση. Τελικά οι Πολωνοί εξέλιξαν το κόμμα αυτό γιατί ήταν η μόνη του ελπίδα που θα έστελνε στη φυλακή την προηγούμενη κυβέρνηση. Πέραν αυτού πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταστραφεί. Ευχαριστώ. Für die fraktion hat jetzt das Wort Herr ο κύριος ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, όταν πριν από δύο χρόνια ανακαλύψαμε το μηχανισμό για το κράτος δικαίου, σε πολλούς δεν άρεσε και αντέδρασαν. Ήταν όμως σημαντικό αυτό και το θέμα δεν είναι η Πολωνία αλλά κάτι πολύ πιο σημαντικό, το κράτος δικαίου, οι, ευρωπαϊκές, οι ευρωπαϊκές κεντρικές σημασίας αξίες. Ίσως σε άλλες χώρες να όφιλε πολύ νωρίτερα να έχει αναλάβει δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως τη Σλοβενία, επί παραδείγματι, όπου ε, η δικαστική εξουσία λειτουργεί πολύ ε, άσχημα, πολλές παραβιάσεις, όπως διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχει γενικώ πολύ κακή εικόνα το δικαστικό σύστημα της Σλοβενίας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι υπάρχει κατάχρηση και παρέμβαση σε πολιτικά θέματα της δικαστικής εξουσίας. Υπήρξε πολιτικός ο οποίος καταδικάστηκε σε επταετή φυλάκιση χωρίς καμία βάση κατηγορίας και ναι μεν ακυρώθηκε μετά η καταδίκη αυτή αλλά η πολιτική ζημιά είχε ήδη γίνει. Η αστυνομία πρόσφατα εισέβαλε στις ε, εγκαταστάσεις, στα γραφεία του μεγαλύτερου κόμματος της ε, αντιπολίτευσης και κατέστρεψε πολλά πράγματα μεταξύ των οποίων και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αντέδρασε σε αυτό. Εγκλήματα δηλαδή και αδικήματα που έχουν διαπράξει άνθρωποι που ανήκουν στο παλαιό καθεστώς. Το ζήτημα λοιπόν είναι, όπως είπα, το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ. Εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών, κυρία Φαϊόν. Tudi Κύριε Πρόεδρε, δεν έχω καμία πρόθεση, κυρία Πρωθυπουργέ, να, κατα... να κατηγορήσω την Πολωνία ή την πολωνική κυβέρνηση. Αντιθέτως, τα τελευταία 30 χρόνια υπήρξε πηγή έμπνευσης για εκατομμύρια Ευρωπαίων η Πολωνία. Μια πολιτική επιτυχία, μια οικονομική επιτυχία χαρακτηρίζει την ιστορία της. Και βλέπουμε ότι έρχεται η ώρα που πρέπει να συζητήσουμε θέματα ε, που μπορεί να απειλούν τις βασικές αξίες. Οι τελευταίες προτάσεις πολωνικής κυβέρνησης μας ανησυχούν ιδιαίτερα. Εγώ ήμουν δημοσιογράφος. Η νομοθεσία αυτή για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποτελεί οξυδρόμη σε σχέση με τις εγγύσεις ανεξαρτησία τους. Εσείς βέβαια ισχυρίζεστε κάτι διαφορετικό παραθέτετε διάφορες οργανώσεις ε, δημοσιογράφων και λέτε ότι θέλετε να ορίσετε μέτρα και σταθμά και νομοθεσία που θα εξασφαλίζει ανεξαρτησία. Πρέπει να μπορεί να γίνει όμως διάλογος και να αναζητηθούν λύσεις. Η Επιτροπή δεν πρέπει να φοβηθεί να επιβάλλει μέτρα όταν υπάρχουν προβλήματα κράτους δικαίου. Είτε πρόκειται για την Πολωνία, είτε για την Ουγγαρία, είτε για τη Σλοβενία ή οποιοδήποτε άλλο κράτος. Λεγκούτκο, συντηρητικοί μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, τέσσερα ζητήματα θέλω να θίξω. Το ένα είναι η γλώσσα. Σημειώνω με ιδιαίτερη ικανοποίηση τον τόνο και το ύφος εντός του οποίου διεξαγάγεται όλη αυτή η συζήτηση και τις εκφράσεις που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής. Ε, το ύφος της Πρωθυπουργού ήταν τόσο πιστικό που ακόμη και ο κύριος Φερχόφστατ νομίζω ότι συμφώνησε με όσα είπατε και πίστηκε. Και αυτό πραγματικά με κατευχαρίστησε. Όμως, να πω αυτό του είδους το ύφος, αυτού του είδους η έκφραση πρέπει να διατηρηθεί. Αυτό που έχουμε δει να συμβαίνει ως τώρα είναι οι λεκτικές επιθέσεις κατά της πολωνικής κυβέρνησης προτού καν αναλάβει καθήκοντα. Αυτό νομίζω ότι είναι παγκόσμιο ρεκόρ σε κάτι που δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Υπόθηκαν ε, πράγματα τα οποία στρεβλώνουν τελείως την επικοινωνία. Εάν μιλά κανείς για πραξικόπημα στην Πολωνία, τότε ή δεν ξέρει γιατί μιλάει ή η θελημενα παραποιεί την πραγματικότητα και χρησιμοποιεί στρεβλές εκφράσεις. Το άλλο στοιχείο είναι τα γεγονότα τα ίδια. Ε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διάβασα ένα έγγραφο που εμφανίστηκε την παραμονή μιας συνεδρίασης του Κολεγίου των Επιτρόπων. Ε, δεν ήρθε από το πουθενά το έγγραφο αυτό. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξή. Πού βρίσκεται αποδεκτικά τη στοιχεία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ποιο σα κάνει αυτέ τι νομικέ αναλύσει και ποιο σας δίνει την επισκόπηση των γεγονότων. Διότι η δική σας παρουσίαση των γεγονότων με αφήνει άναυδο. Παρά τις πληροφορίες που έχει δώσει η πολωνική κυβέρνηση, ε, δεν αναφέρεται καν αυτή η κίνησή της ε, στο συγκεκριμένο έγγραφο. Τις έχετε λάβει αυτές τις απαντήσεις, έχετε πάρει τα στοιχεία και τα αποδεκτικά σας ε, επιχειρήματα ε, του κειμένου αυτού από του ίδιου του εκπροσώπου των μέσων μερική ενημέρωση. Γιατί συντάσσονται αυτά τα έγγραφα. Σα παρακαλώ, κύριοι, πρέπει να παραδεχτούμε ότι τα γεγονότα που αναφέρετε είναι τουλάχιστον αναλυθεί. Το τρίτο ζήτημα είναι τα διπλά μέτρα και σταθμά. Ένα ε, πρόβλημα διαρκείας. Ε, και είναι μια ασθένεια από την οποία νοσεί εδώ και καιρό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κ. Πιτέλε, η κυρία Χάιμς έκαναν λόγο για διαδηλώσεις ήταν στο πλευρό των διαδηλωτών λένε τα περασμένα 8 χρόνια είδαμε πολύ μεγαλύτερες διαδηλώσεις να οργανώνονται στην Πολωνία για άλλα θέματα και Παρόλα αυτά, ούτε η κυρία Χάρμς, ούτε ο κύριος Πιτέλα ε, έχησαν δάκρυα συμπαράστασης για αυτές τις μεγάλες πορείες. Ούτε καν ε, στο κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες δεν πήραν τον λόγο για να μιλήσουν για το θέμα αυτό. Τους μιλήσατε, τους απευθυνθήκατε, μπορεί και αυτοί να είχαν κάτι πολύ σημαντικό να πούνε ε, κυρίες και κύριοι. Συνάδελφοι, τα περασμένα 8 χρόνια στην Πολωνία και αυτό για σας θα πρέπει να είναι μία ε, πληροφορία, μια είδηση που να σημειωθεί. Υπήρχε ένα κράτος μονοκομματικό. Η Πολωνία ε, είχε μόνο ένα κόμμα, ένα πολιτικό κόμμα, το οποίο έκανε κουμάντο σε όλα τα θεσμικά επίπεδα. Και τώρα εξέφνης έχω βρεθεί εδώ και ακούω ότι ε, είναι, ε, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Εάν το δικό μου το κόμμα είχε διορίσει 14 από τους 15 δικαστές στο δικαστηρίο, εδώ θα είχε γίνει ολόκληρη επανάσταση. Πού ακούσατε ότι η, εθνική, η κρατική λαδοτηλεόραση απολύει δημοσιογράφους και υπάρχει λογοκρισία. Κυρίες και κύριοι, αυτή τη στιγμή ε, όλοι σας έχετε παραπλανηθεί τελείως διότι ακούτε αυτά που θέλατε. Προηγουμένω όλοι οι δημοσιογράφοι είχαν απολυθεί από την κρατική ραδιοτηλεόραση και εδώ τι είχε γίνει. Απόλυτη σιωπή, σιγή θύος Διπλά μέτρα και σταθμά λοιπόν. Αυτό αποδεικνύει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρε που είναι πιο ίσε από άλλε. Και υπάρχουν πολιτικά κόμματα πιο ίσα από άλλα. Εάν συνεχίσουμε λοιπόν σε αυτήν την πορεία θα εκτροχιαστούμε. Όχι εμεί οι ίδιοι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η δράση αυτή που αναλαμβάνεται είναι τελείω εναντίον τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Αυτό επίση που θα ήθελα να σχολιάσω ω τελευταίο είναι κάποιοι που ξεπερνούν τα όρια των αρμοδιοτήτων του, των καθηκόντων τους. Κύριε Πρόεδρε, θα ξέρετε ότι το εργαλείο που πάτε να χρησιμοποιήσετε είναι αν μη τι άλλο ύποπτο. Οι νομικές υπηρεσίες των θεσμικών οργάνων το έχουν αμφισβητήσει, δεν θεμελιώνεται ξεκάθαρα στις συνθήκες και είναι πολύ ανησυχητικό από τη νομική οπτική γωνία. Μέλη του Κοινοβουλίου σκοπεύουν να καταθέσουν ψήφισμα, σχέδιο ψηφίσματος σχετικά με το θέμα αυτό και εξ όσων γνωρίζω αναμοχλεύει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά αποδεκτικά στοιχεία με τα γεγονότα πως αναλύονται τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γιατί, γιατί δεν ε, κοιτάζεται το ψήφισμα αυτό να εκπονηθεί ε, στον αέρα. Δεν υπερβαίνετε απλώς το πεδίο των αρμοδιοτήτων σας εσείς. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα υπαγορεύσει ε, τι είδους πλειοψηφία θα πρέπει να απαιτείται στο πολωνικό συνταγματικό δικαστήριο. Αυτό που ε, είπατε δείχνει ότι θέλετε να υπάρξει ένα προηγούμενο. Θέλετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποκτήσει αυτές τις εξουσίες καταχρηστικά, εξουσίες που τώρα δεν έχετε και θέλετε αυτό το εργαλείο να μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και να το εκμεταλλευτείτε για να δράσετε παράνομα και στο μέλλον. Και αυτό είναι το πλέον ανισχυτικό. Για τους φιλελεύθερους η κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Πρωθυπουργέ και εσείς που υποστηρίζετε την κυβέρνηση. Πράγμα το οποίο δείχνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί και τον χώρο συζήτησης των κοινών μας αξιών. Δεν πρόκειται για εθνικά θέματα, δεν πρόκειται για επίθεση στη μία ή στην άλλη χώρα, πρόκειται για τις ίδιες τις αξίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Τώρα η πολωνική κυβέρνηση με την πλειοψηφία με την οποία κέρδισε έχει την ευθύνη να μεγιστοποιήσει το χώρο και όχι να τον ελαχιστοποιήσει για κριτική. Πρέπει να ενισχύσετε τις οροπίες και του ελέγχους, όχι να τα αποδυναμώσετε. Δεν ξέρω αν ακούσατε προσεκτικά, αλλά εγώ δεν είμαι σίγουρη ότι πρέπει να πάρετε σαν παράδειγμα τον κύριο Ορμπάν ή δεν ξέρω ποιον άλλον τον Πούτιν. Πιστεύω λοιπόν ότι η πρωτοβουλία της Επιτροπής δικαιολογείται δεν πρέπει να την κατηγορείτε ότι μεροληπτή. Βέβαια εντάξει μπορούμε να πούμε γιατί Πολωνία και όχι Ουγγαρία. Η συζήτηση πάντως εδώ σήμερα δείχνει ότι χρειάζεται ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός που να βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια με διαφάνεια για να αξιολογούνται όλες οι χώρες μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με τον ίδιο τρόπο. Βλέπω ότι χαμογελάει ο κύριος Τίμερμαν, γιατί ξέρει ότι εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετοιμάζουμε ένα τέτοιο μηχανισμό. Κύριε Τίμερμαν, κύριε Κούντερς, αν το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεχτεί την πρόσκληση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπονήσουν ένα τέτοιο μηχανισμό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Σπινέλη τώρα εκ μέρου τη ΓΚΟΕ, παρακαλώ. Θα συμμεριστώ τις ανησυχίες πολλών από τους συναδελφούς. Ο, ο νέο εθνικισμός ε, της κυβέρνησής σας, ε, κυρία Τζίτλο, ε, οι περιορισμοί που έχετε προβλέψει και περιορίζουν τις εξουσίες του Συνταγματικού Δικαστηρίου και τις ελευθερίες των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλα αυτά αντίκεινται στην αρχή της ευρωπαϊκής σας κατεύθυνση. Εάν η Πολωνία ενέκρινε μια κυβέρνηση που επικρίνει τόσο πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση, βέβαια, είναι επειδή με τι πολιτικέ λιτότητά τη η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε σε αυτή τη χώρα ανισότητε πάρα πολύ οξυμένε και κοινωνικές αδικίες που μόνο η δεξιά ξέρει να εκμεταλλεύεται τόσο επάξια. Ακόμη και η κοινωνική δικαιοσύνη είναι ένα ευρωπαϊκό δικαίωμα. Θα πρέπει όμως να μην χρησιμοποιούνται διαφορετικά κριτήρια στην Ουγγαρία και την Πολωνία ή όπως έγινε χθε στην Ιταλία. Τις κυβερνήσεις πρέπει να τις αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο ισότιμο τρόπο. Η Πολωνία δεν μπορεί να, καταβάλει ψηλότερο τίμημα μόνο και μόνο γιατί η κυβέρνηση της ε, έχει αναλυθεί από ε, μια, από ένα κόμμα λιγότερο ισχυρό από το ΕΛΚ, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστούμε και τώρα η κυρία Σαρχεντίνη για τους πρασίνους. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Πρόεδρε, μην έχουμε αμφιβολίες για το τι συμβαίνει όσον αφορά τις αποφάσεις της ε, Πολωνικής και την αντιδημοκρατική τάση. Εγώ θέλω να μιλήσω κυρίως για τον Υπουργό Εξωτερικών της Ολλανδίας, και για το τι κάνουμε εμείς με τις γείτονες χώρες, για τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η αξιοπιστία, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Τίμερμανς. North Stream λοιπόν, ο αγωγός αυτός, η Πολωνία αρνήθηκε, φοβάται τη Ρωσία. Είναι λογική η πολιτική αυτή, κύριε Κούντερς. Και η Πολωνία ενισχύει τις απόψεις του κύριου Βίλντερς. Ο Πρωθυπουργός Ρούιτε, Πρωθυπουργός της Ολλανδίας, δεν αποστασιοποιείται. Και προσκλήθηκε η Πρωθυπουργός να έρθει εδώ να μας ενημερώσει. Οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης δεν ικανοποιούνται από αυτή τη διαδικασία. Όλα αυτά δεν οδηγούν σε αξιοπιστία κυρία Πρωθυπουργέ. Πρόεδρε, εδώ πρέπει να πάρουμε μαθήματα. Και μόνο αφού πάρουμε εμείς μαθήματα θα μπορούμε και εμείς για αυτά τα ευαίσθητα θέματα να μιλάμε. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του FTD, ΜΑΧ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αντιμετωπίζουμε μια σκανδαλώδη κατάσταση σήμερα, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει μια διαδικασία σε βάρος της Πολωνίας, που μπορεί να καταλήξει στην απόσυρση του δικαιώματος ψήφου της Πολωνίας. Και γιατί, γιατί αποφάσισε να ισχύσει η πλειοψηφία των δύο τρίτων στο συνταγματικό δικαστήριο και να αλλάξει την κατάσταση όσον αφορά τα μέσα ενημέρωση. Μα είναι μια συνηθισμένη αυτή η κατάσταση και σε άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για πρόσχημα. Τι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα δεν της αρέσει που κέρδισε ένα κόμμα που δεν υποστηρίζει έθερμα την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ότι κέρδισε τις εκλογές, αυτό την ενοχλεί, το ότι δεν θέλει να εφαρμόσει τις ποσοστώσεις για τη μετανάστευση. Όντως περί αυτού πρόκειται. Τίποτα άλλο δεν έχουμε να κάνουμε εδώ πέρα παρά την ανάμειξη στα εσωτερικά μιας κυρίαρχης χώρας. Ο το 1963 στο δυτικό Βερολίνο είπε το περίφημο «Είμαι Βερολινέζος». Σήμερα λοιπόν πρέπει να είμαστε με την Πολωνία, η οποία αποτελεί θύμα άδικων επιθέσεων από πλευρά της Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θα πω και εγώ, ναι, είμαι Πολωνός. E Ευχαριστούμε για την ΕΝΕΦ, e ο κύριος Σοφοζέρ. Κυρία Πρωθυπουργέ, ε, αγαπητοί συνάδελφοι, ο κύριος Σούλτ μίλησε για παρεξικόπημα και για πουτινοποίηση της πολωνικής ε, πολιτικής. Κι όμως ε, το PIS, το κόμμα δικαιοσύνης και νόμου της Πολωνίας, είναι ένα δημοκρατικό κόμμα. Μιλάμε για επίθεση κατά της δημοκρατίας και της εθνικής κυριαρχίας της Πολωνίας εδώ. Η ελευθερία και η ανεξαρτησία μέσα στην ελληνική είναι δικαίωμα του πολωνικού λαού και όλοι οι λαοί της Ευρώπης πιστεύουν στις αρχές του ανθρωπισμού. Στον ανθρωπισμό δεν προβλέπεται κατασκευή μιας νέας τάξης της Ευρώπης που θα καταργεί το δικαιώματα και την πραγματική τάξη. Οι Πολωνοί έχουν αντισταθεί μετά την πτήση του τείχους και αντιστέκονται ακόμη διότι ε, είναι μια χώρα συντηρητική, αρχαία και αληθινή. Θα πρέπει λοιπόν το σεβασμό της ζωής την αλήθεια, τα δικαιώματα, τη δικαιοσύνη, την καθηλική θρησκεία και όχι τον νεοφιλελευθερισμό όσων μάχονται την κοινωνία με τα οικονομικά μέσα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να τα αφήσουμε ανεξέλεκτα. Η Ευρώπη είναι μια αποτυχία, είναι μια δικτατορία που υποχρεώνει τους λαούς να υποκληθούν μπροστά στις επιταγές μιας συνθήκης και, ε, να, ε, και φημώνει όσους τολμούν να καταψηφίσουν το ευρωπαϊκό σύστημα. Το ευρωπαϊκό, ε, το ευρωπαϊκό σύστημα ε, πλήττει τις χώρες, ε, την Πολωνία, την Τουρκία, όλες αυτές τις χώρες που αντιστέκονται κατά αυτής της δικτατορίας που είχαν κάνει τη βελούδινη επανάστασή του στο παρελθόν και την οποία σέβομαι και χαιρετίζω, που δεν θέλουν να υποκληθούν σε αυτά τα ξένα συμφέροντα που κάνουν κουμάντο εδώ και ποδηγετούν τους ευρωπαϊκούς λαούς. Θα πρέπει να αντισταθούμε και στη γερμανική αλαζονία. Εμείς οι Γάλλοι είμαστε στο πλευρό της Πολωνίας και δεν μπορούμε να δεχτούμε η Γερμανία ε, να καθορίζει το τι θα συμβεί στην Ευρωζώνη και να θυμώνει την ε, ευρωπαϊκή ε, τόλμη και ζωτική ενέργεια. Η Πολωνία είναι μια χώρα κοινωνικού συντηρητισμού, χριστιανική χώρα και δημοκρατική. Εδώ λοιπόν η επανάσταση των λαών έχει αρχίσει, σας προειδοποιώ. Και αυτά που αξίζετε θα τα πάρετε. Η ώρα πλησιάζει. Ich muss das jetzt leider noch mal wiederholen, meine Damen und Herren auf den Tribünen. Äh, θα επαναλάβω κυρίες και κύριοι ότι απαγορεύεται ρητά από τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εκδηλώνεται χειροκροτήματα ή αποδοκιμασίες. Σας φιλοξενούμε εδώ, αλλά είμαι βέβαιος ότι στο Πολωνικό Κοινοβούλιο τα πέντε λεπτά δεν θα σας άφηναν στις εξέδρες εάν παραβιάζετε τον κανονισμό. Γι' αυτό παρακαλώ να απέχετε από οποιαδήποτε επίδειξη, εκδήλωση ε, προτίμηση. Ο κύριο Σοφχάτ. Κυρία Πρωθυπουργέ, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ακούω την κυρία Χάμπ, τον κύριο Φερχόφστατ να μιλάνε, αλλά διαπιστώ και διαπιστώνω ότι το πρόβλημα δεν το έχει με το κράτο δικαίου η Πολωνία. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα έχουν πρόβλημα με τη δημοκρατία και το κράτο δικαίου. Όταν ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιλάει για το υποτιθέμενο πρόβλημα τη ε, Πολωνία, Διαπιστώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πρόβλημα προ την πραγματικότητα, τα γεγονότα. Έχει κοιτάξει ποιο ήταν ο χρόνο ομιλία, πριν από την εκλογή του κόμματο δικαίου και δικαιοσύνη, ε, του χρόνου μιλία που διατίθεται στι διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις, τον τρόπο λειτουργία ε, των δικαστηρίων. Θεωρείτε ότι ο πολιτικός λαός, ο οποίος αγωνίστηκε για την ελευθερία του, είναι διατεθειμένος να την παραδώσει έτσι. Ο Πιότρ Καζίνσκι, πολιτιολόγος Πολωνός, που άλλωστε δεν είναι και πολύ γνωστό, δεν θεωρείται ε, υποστηρικτής του κόμματος Δίκαιο και Δικαιοσύνη. Το διάβασα πρόσφατα. Λέει ότι δεν υπάρχει ε, παρεκτροπή προς το φασισμό στην Πολωνία. Επιθυμίζω ότι τα μέλη του Συνταγματικού Συμβουλίου στην πατρίδα μου τη Γαλλία εκλέγονται άμεσα και έμεσα αντίστοιχα του Ροδιατηλεοπτικού Συμβουλίου από τον ε, πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Γερουσίας και της ε, Γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να θεωρηθεί ως μια έμεση επέμβαση της πολιτικής εξουσίας. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι υπάρχουν ε, εδώ προσχήματα τα οποία αξιοποιούνται για να αποσταθεροποιηθεί μια κυβέρνηση και δύο πολωνική. Και εγώ δηλώνω εδώ με παρησία είμαι Πολωνός, ο Πρόεδρος διακόπτη. Εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο κύριος Ολμπριχτ. Ευχαριστώ πολύ, Πρωθυπουργέ, κυρίες και κύριοι. Η Πολωνία είναι ένα κοινό αγαθό του συνόλου των πολιτών της και θα πρέπει να τη φροντίσουμε. Είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα μας και είμαστε υπερήφανοι για την δράση των Πολωνών οι οποίοι έχουν θεωρηθεί πολλές φορές πρότυπα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραδείγματα για την υπόλοιπη Ευρώπη, ανεξαρτήτως της τάσης της κυβέρνησης της χώρας. Λυπούμεθα που η Πολωνία είναι το θέμα μια συζήτησης για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει για τη χώρα μου και ελπίζω να είναι και η τελευταία. Γνωρίζετε ότι δεν προκαλέσαμε εμείς Πρωθυπουργέ τη συζήτηση αυτή. Εμείς προσπαθήσαμε να την αποτρέψουμε τη συζήτηση αυτή. Παρ' όλα αυτά η συζήτηση θα επηρεάσει την εικόνα της χώρας σε διεθνές επίπεδο. Γνωρίζουμε ότι κερδίσατε τις τελευταίες εκλογές στην χώρα σας, στη χώρα μας μάλλον, δεν αμφισβητούμε την εκλογική σας νίκη και δεν αμφισβητούμε το δικαίωμά σας να εφαρμόζετε ένα πολιτικό πρόβλημα το οποίο να διαφοροποιείται από το δικό μας. Αυτό σημαίνει ότι ε, έχετε τον έλεγχο φυσικά της χώρας, ελέγχετε τις υπεύθυνε θέσεις, είστε όμως και υπεύθυνοι και υπόλογοι για όλες τις αλλαγές οι οποίες μπορεί να συμβούν σε επίπεδο κρυθμίσεων κράτους δικαίου. Νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει βλάπτει την εικόνα της χώρας στην Πολωνία και στον κόσμο. Λοιπόν, είστε υπεύθυνοι για τη συζήτηση αυτή πλέον, διότι είστε Πρωθυπουργό. Η Πολωνία πάντως δεν συνηθίζει να προκαλεί τις υπόλοιπες χώρες με τέτοιο τρόπο και αυτό μας λυπεί. Ο κύριος Βάιντεν Χόλτσα έχει το λόγο εκ μέρους των Σοσιαλδημοκρατών. Παρακαλώ να ανοίξετε και το μικρόφωνο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Πρωθυπουργέ. Χαιρετίζω τη σημερινή συζήτηση και το γεγονός ε, ότι διεξάγεται σήμερα και το γεγονός επίσης ότι διεξάγεται και επί της ουσίας. Δεν πρόκειται για την καταδίκη της ε, Πολωνίας. Η Πολωνία είναι μια πολύ σημαντική χώρα που άφησε το στίγμα τη στην ευρωπαϊκή ιστορία. Οι Πολωνοί συνέβαλαν τα μάλα στην αντιμετώπιση της ε, κομμουνιστικής δικτατορίας. Η Ευρώπη χωρίς ε, την Πολωνία ε, θα ήταν ατελής. Εμείς σεβόμαστε την ψηφοφορία, την ψήφο του πολωνικού λαού, αλλά ξέρετε ανησυχούμε πάρα πολύ γιατί τα μέτρα που λαμβάνει η πολωνική κυβέρνηση δημιουργούν κάποιο φόβο στους Πολωνούς. Βεβαίως και η αλλαγή είναι αδιαμφισβήτητη αρχή της εξουσίας, αλλά αυτό δεν πρέπει να οδηγεί στο να αλλάζουν οι κανόνες με τέτοιο τρόπο που να μην μπορούν να βελτιωθούν στο μέλλον. Αυτό φοβούνται οι περισσότεροι Πολωνοί. Τα μέτρα που λήφθησαν στον τομέα της ε, δικαιοσύνης έχουν τροφοδοτήσει αυτό το φόβο. Ε, ο σεβασμός ε, των μειονοτήτων είναι επίσης μια διαμφισβήτητη αρχή της δημοκρατίας. Και σε αυτό το θέμα υπάρχουν πάρα πολλές σχετικές διαμαρτυρίες. Η Πολωνία είναι εκείνη που μας χάρισε το θεσμό της στρογγυλής τράπεζας και θέλω να επενθυμίσω στην κυβέρνηση ότι ο διάλογος είναι καθοριστική σημασία. Είναι πολύ σημαντικό το ότι διεξάγεται σήμερα συζήτηση εδώ, να ξεκαθαριστεί η κατάσταση, να μην υπάρχουν πλέον αμφιβολίες. Η συζήτηση πρέπει να διεξαχθεί με ανοιχτό τρόπο άμεσα, γιατί με τον τρόπο αυτό και η Πολωνία θα κερδίσει αλλά και η Ευρώπη. Πολύ ωραία. Ο κύριος Χένκελ εκ μέρους του ECR. Καταρχήν, κύριε Πρωθυπουργέ, ε, ήθελα να σας εκδηλώσω το σεβασμό μου για το ότι κάθεστε εδώ και ακούτε η ίδια αυτή την κατά κάποιον τρόπο παράδοξη ιερά εξέταση. Κύριε Βάινχολτσε, πολύ σωστά επισημάνατε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καταδίκη εκ των προτέρων. Μόνο που πρέπει να ρωτήσω τον ε, πρόεδρο του Κοινοβουλίου τι εννοεί Πώς το εννοεί ότι η δημοκρατία, μάλλον η Πολωνία, είναι δημοκρατία ε, όπως την εννοεί ο Πούτιν. Δεν είναι αυτό εκ των προτέρων καταδίκη. Κύριε Σούλτς, πρέπει να σας πω, εγώ ε, πολλές φορές έτρεξα πολύ γρήγορα και οποτεδήποτε με συνέλαβαν, ζήτησα συγγνώμη. Μήπω θα πρέπει κύριε Σούλτ και εσεί σήμερα εδώ να ζητήσετε συγγνώμη. Δεν νομίζετε ότι προσφέρετε ευκαιρία για να ζητήσετε συγγνώμη. Ο καθηγητής Λουκ επισήμανε ότι δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και εγώ αυτό πρεσβεύω. Και θα σας αναφέρω και κάποια άλλα παραδείγματα για τη διακριτική μεταχείριση. Πιστεύω η Πολωνία αντί να ασχολείται, μάλλον η Κομισιόν αντί να ασχολείται με την Πολωνία, να ασχολείται καλύτερα με τις ε, διαδικασίες επιπαραβάση των ε, ευρωπαϊκών θεσμών ή των μεγάλων χωρών. Και θέλω να πω, υπάρχουν πάρα πολλές παραβιάσεις της συνθήκης του Μάστριχτ από την Ευρωζώνη. Ή ο κανόνας ε, της ε, αγοράς ε, αποβλήτων από την ΕΤΣΕΠΕ ή η παραβίαση του συμφώνου του Δουβλίνου από την καγκελάριο κυρία Μέρκελ. Γιατί λοιπόν η Κομισιόν ενδιαφέρεται για το πολωνικό συνταγματικό δικαστήριο αλλά όχι για το ότι τρεις πρώην δικαστές του γερμανικού συνταγματικού δικαστηρίου αποφάρθηκαν και είπαν ότι η πολιτική προσφύγων της Γερμανίας είναι αντισυνταγματική γιατί δεν ενδιαφέρεστε γι' αυτό. Κύριε Oettinger, επίσης θα πρέπει λιγάκι να εξτάσετε το εξή ερώτημα. Η ε, κρατική τηλεόραση της Γερμανίας που χρηματοδοτείται με χρήματα των Γερμανών. Μήνες ολόκληρους ε, παρουσιάζει το προσφυγικό με αισιόδοξα χρώματα, ωραία χρώματα και αγνοεί το τι συμβαίνει με τη συμπεριφορά των Βόρειο Αφρικανών. Κυρίες και κύριοι, οι Γερμανοί οφείλουν την πτώση του τείχους, του στην Πολωνία. Και υπενθυμίζω την περίπτωση Σολιντερνόσκ, ε, κάποια μέλη της ολυνταρνό και βρίσκονται σήμερα σε ηγετικέ θέσεις της πολωνικής κυβέρνησης. Στην αρχή οι Γερμανοί πολιτικοί ήθελαν να σώσουν ε, το κλίμα μετά το ευρώ τρεις φορές στην Ελλάδα, τους πρόσφυγες και τώρα θέλουν να σώσουν και την πολωνική δημοκρατία. Κυρίες και κύριοι, αν ένας λαός δεν χρειάζεται καμία βοήθεια, δεν χρειάζεται να κάνει ιδιαίτερα μαθήματα για τη δημοκρατία, αυτός ο λαός είναι η Πολωνία. Τώρα, η κυρία Βίξτρομ από τους ε, φιλελευθέρους. Ευχαριστώ κύριε ε, Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής ευθύς εξ αρχής και να πω ότι ακόμα και αν επικρίνουμε τα ε, όσα σήμερα συμβαίνουν στην Πολωνία θα πρέπει να τονίσουμε ότι θα πρέπει πάντα να είμαστε σε θέση να συζητούμε ειλικρινά μεταξύ μας και παρόλα αυτά να παραμένουμε φίλοι, παρόλες τι απόψει που μπορεί να διαφέρουν. Η Πολωνία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κράτος στην Ευρώπη. Τα βασικά θεμελιώδη δικαιώματα θα πρέπει να προστατεύονται σε οποιαδήποτε χώρα της Ένωσης. Κύριε Επίτροπε Τίμερμανς, ε, είναι πολύ σωστό αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάζει τα τεκτενόμενα στην Πολωνία, αλλά υπάρχει και μια υποκρισία εδώ. Ή θα ήταν υποκρισία εάν δεν κοιτούσαμε τι συμβαίνει ταυτόχρονα στην Ουγγαρία. Είναι φυσιολογικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παρακολουθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη θεμελιώδη και το κράτος δικαίου σε όλα τα κράτη-μέλη με τον ίδιο τρόπο. Κυρία Πρωθυπουργέ, αν συνεχίσετε σε αυτή την ατραπό υπάρχει ένας κίνδυνος να υπονομεύσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις εμελιώδεις ελευθερίες και στη χώρα σας και αλλού. Δεν θέλουμε να δούμε ντόμινο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία χώρα να παρασύρει την επόμενη ε, ε, στην κατηφόρα αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντίθετα, εμείς θα πρέπει να αντισταθούμε και να προστατεύσουμε τις αρχές και τις αξίες μας. Αυτά είναι τα ίδια τα θεμέλια για το τεράστιο εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό θα χρειαστούν οι επόμενες γενναίε. Ευχαριστώ. Από ε, την Ενωτική Αριστερά το λόγο έχει ο κύριος Λουιέρικ. Αν κατάλαβα καλά τις εξηγήσεις οι οποίες μας δόθηκαν, μειώνουμε τη δημοκρατία για να την ενισχύσουμε. Η Πολωνία ζητά να εξαιρεθεί από τη χάρτα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στο όνομα της βελτίωσης του σεβασμού των δικαιωμάτων αυτών. Τι πίστη να δώσουμε στη συζήτηση η οποία γίνεται σήμερα όταν τα θεσμικά όργα αποφάσισαν να δωρήσουν 3 δις ευρώ στην Τουρκία του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος και αυτό διώκει τους δημοσιογράφους, τους φυλακίζει και ελέγχει τη δικαιοσύνη. Η Ευρώπη της αγοράς έχει υποκαταστήσει την Ευρώπη της ελευθερίας, των αρχών, των δημοκρατικών δικαιωμάτων, του πλουραλισμού. Εγώ θα έλεγα να υπάρξει ένας ειδικό επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που να ασχολείται με τα θέματα αυτά σε κάθε χώρα. Δεν είναι αργά. Ε, ένα τέτοιο παρατηρητήριο θα μπορούσε να ελέγχει επίσης και τη λειτουργία των μέσων τήρησης και σεβασμού του δικαίου στις διάφορες χώρες. Ευχαριστώ από τους Πρασίνους, ο κύριος Κάμπρας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Πρωθυπουργέ, μιλώ ως Πρόεδρος της ε, Ομάδας για την Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία στο Κοινοβούλιο. Το 2011 στην τελευταία απογραφή 847.000 ε, άνθρωποι δήλωσαν ότι είναι από τη Σιλεσία. Μόλις πριν από τέσσερις μέρες ο Γέρση Μπούσελικ εξ ονόματος 140.000 ζήτησε να αναγνωριστεί ε, η εθνική μειονότητα ε, της Σιλεσίας στην Πολωνία, των Σιλεσιανών ενώ το κυβερνών κόμμα και οι βουλευτές του τους απείλησαν με διώξεις, ακόμα και εκτελέσεις. Ακόμα δεν καταγράφονται ως εθνική μειονότητα, ούτε αναγνωρίζεται η περιφερειακή τους γλώσσα σύμφωνα με ε, ε, το κατάλογο του 2005. Είναι μια κατάσταση που μας έχει θορυβήσει και μας δημιουργεί αγωνίες. Τι γίνεται εκεί ε, με την καταστολή των μειονοτήτων στην Πολωνία αυτό θα ήταν και αντιδημοκρατικό και επέσχυντο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Τερικάβρας. Από την ΕΝΕΦ το λόγο έχει ο κύριος Μπέ από την Ευρώπη της ε, Ελευθερίας. Πρωθυπουργέ, μετά τον Βικτόρ Ορμπάν είναι η σειρά σας να έρθετε εδώ για να απαντήσετε στις σκανδαλώδεις κατηγορίες τη βάρος της κυβέρνησής σας από πλευράς της Ευρωκρατία κατηγορήστε ότι εφαρμόζετε το πρόγραμμα, το προεκλογικό, το οποίο σας οδήγησε στην εξουσία με εντελώς δημοκρατικές εκλογές. Εσείς προσπαθείτε να προστατεύσετε τους Πολωνούς από τις παράλογες αποφάσεις των Βρυξελών στον τομέα της μετανάστευσης. Εσείς αντί να κάνετε έκκληση για περισσότερους μετανάστες βοηθάτε τις οικογένειες της Πολωνίας που βοηθάτε με 500 λότια ανά παιδί. Μετά από την ταραχώδη συζήτηση που προηγήθηκε, θα ήθελα να πω ότι σας ευχαριστώ γιατί δείξατε ότι μια άλλη Ευρώπη είναι εφικτή. Μια ελεύθερη κυρίαρχη Ευρώπη με ελεύθερους κυρίαρχους λαούς. Βλέπω ότι με χαρά μαζί με τους Ούγκρους, τους Τσέχους και τους Σλοβάκους δημιουργείται ένα ομοιογενές μπλοκ που αρνείται της, ε, Ευρωπαγκοσ... της δυνάμεις της ευρωπαγκοσμιοποίησης. Ζήτω η ελεύθερη και περήφανοι λαοί. Λοιπόν, το λόγο έχει τώρα η Πρωθυπουργό της Πολωνίας, η κυρία Σίτλο, παρακαλώ. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για όλες τις παρεμβάσεις και τα καλά σας λόγια και τα λόγια υποστήριξης, ακόμα και τα λόγια ανησυχία που εκφράσατε. Νομίζω ένα πράγμα μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Ανησυχούμε βαθύτατα και νοιαζόμαστε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τη μελλοντική της μορφή. Εμείς όλοι θέλουμε και η Πολωνία θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ε, ε, σταθερή δεν θέλουμε ε, να ε, ταράσετε και να μαστίζεται από κρίσεις η Ευρώπη. Η Πολωνία δεν ευθύνεται για τις κρίσεις αυτές και θέλει να είναι ε, πρωταγωνιστής στη διαμόρφωση ευρωπαϊκών πολιτικών τέτοιων που θα μας επιτρέψουν να αποτρέπουμε μελλοντικά προβλήματα. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για την υποστήριξη και για τις επικρίσεις ακόμα που εκφράζετε. και σας ευχαριστώ για την υποστήριξη για τη χώρα μου και την κυβέρνησή μου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας και ήρθα εδώ να μοιραστώ κάποιες ε, πληροφορίες που έχω μαζί σας και να προσπαθήσω να δράξω την πρώτη ευκαιρία που έχω να σας μιλώ για να σας ενημερώσω σε μεγαλύτερο βάθος ε, για κάποια σημαντικά ζητήματα που σας ανησυχούν από ό,τι βλέπω. Ε, το ένα είναι ε, ε, το συνταγματικό δικαστήριο και το άλλο ο νέος νόμος για τα μέσα ενημέρωσης. Περίμενα πιο λεπτομερείς ερωτήσεις να γίνουν για αυτά τα θέματα. Ε, πάντως δεν με ρωτήσατε αυτά που περίμενα. Άρα, μάλλον δεν θα υπάρχουν προβλήματα αν δεν έχετε λόγο να μου κάνετε λεπτομερείς ερωτήσεις. Τι να υποθέσω, Όλη η συζήτηση αυτή είναι για μας πρόβλημα που θα πρέπει εγώ να αντιμετωπίσω προσωπικά και να το λύσω. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θέλει να εφαρμόσει τώρα την ε, απόφαση που έλαβε και να την επιβάλλει στην Πολωνία. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να έχουμε γνώση όλοι των πραγμάτων για να αγωνιζόμαστε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που να λειτουργεί με ε, στιβαρά θεσμικά όργανα και αξιόπιστα και λειτουργικά. Ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε περισσότερο ε, τις αρμοδιότητές μας και τον τρόπο με τον οποίο στο μέλλον εργαζόμαστε. Θα ήθελα να επαναλάβω μερικά σημαντικά στοιχεία που μπορεί να σας διέφυγαν από την πρωτομιλία μου. Νομίζω ότι η Πολωνία πραγματικά δεν αξίζει να υφίσταται την επιτήρηση για την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν υποφέρουν, το κράτος δικαίου δεν παραβιάζεται επίσης και όλη η δουλειά που γίνεται τώρα στην Πολωνία συνάδει απολύτω και με τι ευρωπαϊκέ συνθήκε και με την πολωνική νομοθεσία. Είμαστε κυρίαρχο κράτο. Είμαστε ελεύθερη χώρα. Επιτρέψτε μου παρεμπιπτόντως να σας πω ότι στην Πολωνική Βουλή ε, προσκεκλημένοι και οι θεατές ε, επιτρέπεται να εκφράσουν την επιδοκιμασία τους ή την αποδοκιμασία τους. Αλλά αυτή είναι η δική μας παράδοση. Ε, επιτρέπεται το κοινό δηλαδή να εκφράζεται, να εκφράζει τις απόψεις και τα ε, συναισθήματά του και μας είναι ιδιαίτερα προσφυλής και η ελευθερία μας γιατί έχουμε πληρώσει ένα πάρα πολύ υψηλό τίμημα και θα την υπερασπιστούμε και την έχουμε υπερασπιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας μας. Έχουμε βγάλει και διδάγματα από την ιστορία και τα διδάγματα είναι ότι τα πολωνικά προβλήματα θα πρέπει να συζητιώνται και να λύνονται στην Πολωνία. Γιατί όποτε προσπάθησαν τρίτες δυνάμεις να λύσουν τα προβλήματα για λογαριασμό μας ήταν ολέθριο για την Πολωνία αυτό. Οπότε αυτό λέγω. Δεν λέγω ότι συμφωνούμε όλοι, ούτε θέλω να εμφανίσω μια ψευδή εικόνα. Υπάρχουν διαφωνίες και η διαφωνία ίδια είναι συστατικό της ε, δημοκρατικής συζήτησης. Αλλά η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνει εκεί που αρμόζει, στην Πολωνική Βουλή. Η καλύτερη απόδειξη για το γεγονό ότι είναι δημοκρατική χώρα η Πολωνία είναι η εξής. Σήμερα στη Βουλή έχουμε Πολωνούς πολίτες οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα ε, να εκφράζουν και τις ε, διαφωνίες τους με την κυβέρνηση. Ξέρετε ότι γίνονται και διαδηλώσεις. Είναι δημοκρατική χώρα η Πολωνία και εδώ έχω έρθει ενώπιόν σας ως Πρωθυπουργό μιας δημοκρατικής χώρας. Ανησυχώ βαθύτατα διότι επιθυμώ όλοι να έχουμε ένα κοινό μοντέλο για τη μελλοντική μας συνεργασία και ε, λειτουργία στην Ευρώπη για να αποφεύγονται τέτοιου είδους συζητήσεις. Διότι αυτές δεν έχουν νόημα και δεν έχουν και καμία βάση ουσιαστική οι συζητήσεις. Ήρθα λοιπόν εδώ ενώπιόν σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για έναν ακόμα λόγο. Έχω βαθύτατη αίσθηση της ευθύνης. Όχι μόνο για τον όσων συμβαίνουν σήμερα στην Πολωνία αλλά και στην Ευρώπη εν γέννη Βλέπετε λοιπόν να σας μιλώ για τη μετανάστευση που είναι τεράστιο πρόβλημα και το γνωρίζετε άλλωστε πάρα πολύ καλά. Η Πολωνία ήδη έχει ε, υποδεχτεί πάνω από ένα εκατομμύριο Ουκρανούς. Κανείς δεν τους ήθελε, τους θέλαμε εμείς. Είναι στην Πολωνία και αυτό δεν πρέπει να το συζητήσουμε. Είναι ένα ζήτημα για την πολωνική κυβέρνηση που θέλει να συζητήσει για τη μετανάστευση. Είμαστε μια χώρα που λειτουργεί με βάση το κράτος δικαίου και λαμβάνουμε τις αποφάσεις που έλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση γιατί η χώρα έχει συνέχεια και θα συζητήσουμε και τους μηχανισμούς μετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να το λύσουμε το μεταναστευτικό. Θα πρέπει όλοι να κληθούμε να απαντήσουμε, ιδιαίτερα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι αυτό περιμένουν οι πολίτες της Ευρώπης από εμά και από εσά. Αυτό είναι βασικός στόχος για μας και μεγάλη πρόκληση. Δεν θέλω οι Πολωνοί να γίνουν ευρωσκεπτικιστές. Δεν θέλω οι Πολωνοί να ε, είναι απέναντι στην Ευρώπη, να την αντιμετωπίζουν ε, κριτικά. Γι' αυτό θέλω η Ευρώπη να γίνει μια κοινότητα κρατών κυρίαρχων που να διοικούνται και να κυβερνώνται με σωστό τρόπο. Η ε, κυβέρνηση της Πολωνίας δεν πρόκειται να απεμπολίσει το πρόγραμμά της. Πρόγραμμα με το οποίο επιφορτίστηκε μετά από τις ελεύθερες εκλογές που ήταν και πάρα πολύ πρόσφατες. Κερδίσαμε τις εκλογές ακριβώς βάσει του προγράμματός μας διότι έτσι αποφάσισαν οι Πολωνοί πολίτες. Τώρα, από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε το δικό μας πρόγραμμα. Διότι ο λαός γι' αυτό μας ψήφισε. Οι Πολωνοί έχουν την αίσθηση ότι έχει αδικηθεί η Πολωνία. Θέλουμε ίσες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Εμείς οι Πολωνοί θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός αυτό να μετράμε την επιτυχία μας με γνώμονα τις πιο επιτυχημένες χώρες στην Ευρώπη. Εμείς είμαστε σχετικά νέο μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενταχθήκαμε στην Ένωση κουβαλώντας τη δική μας ιστορία, όπως και άλλες χώρες της Κεντρικής Ευρώπης και Ανατολικής. Αλλά ήρθαμε με πολλές ελπίδες τότε και ήταν θαύμα όνειρο για μας το γεγονός ότι ενταχθήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν το απάβγασμα της ε, ισότητας και της δικαιοσύνης και τέτοια Ευρώπη θέλουμε. Βέβαια τα πράγματα δεν είναι καθόλου εύκολα γιατί παραμένουν κάποια εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουμε αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τα υπερβούμε. Σήμερα αυτό που χρειάζεται η Πολωνία είναι δουλειά για να βελτιώσουμε το κράτος και τη λειτουργία του ο πρόεδρος Καζίνσκι, πρώην πρόεδρος που έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, είπε ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι μια χώρα και για τους αδυνάτους. Ε, αυτή την πρόκληση δεν την έχουμε αντιμετωπίσει, είναι ακόμα μπροστά μας. Όπως και ο μακαριστός ο Πάπας Ιωάννης Παύλος δεύτερος είπε «Μη φοβάστε ποτέ, μη φοβάστε ποτέ λοιπόν, ας είμαστε όλοι υπέρ μια δίκαιη Ευρώπης, μιας ελεύθερης Ευρώπης και α αγωνιστούμε από κοινού γι' αυτό. Ας μην φυσούμε καμία προσπάθεια, κανένα σκόπου, έτσι ώστε όλοι οι Ευρωπαίοι να έχουν την αίσθηση ότι υφίστανται ίση και δίκαιη μεταχείριση. Η Πολωνία δεν αξίζει αυτή την κριτική που δέχεται σήμερα. Επιτρέψτε μου να σας υπενθυμίσω ότι υποχρεωθήκαμε να τροποποιήσουμε τον προηγούμενο νόμο ε, για τη λειτουργία του συνταγματικού δικαστηρίου, διότι η απελθούσα κυβέρνηση αποφάσισε να επιταχύνει ε, τις εργασίες για το συνταγματικό δικαστήριο, τις νομοπαρασκευαστικές. Το 2012 κατέβηκε το πρώτο νομοσχέδιο ε, αλλά στη συνέχεια δεν ακολούθησε καμία ενέργεια. Αποφάσισε λοιπόν το συνταγματικό δικαστήριο ότι ήταν αντισυνταγματικός αυτός ο νόμος, το νομοσχέδιο. Οι δικέ μα θέσει έχουν πλειοψηφία στο συνταγματικό δικαστήριο. Τώρα εσεί αναφερθήκατε και στα μέσα ενημέρωση. Πώ στείνουμε το μηντιακό μα σύστημα, όπω και στην Ιταλία για παράδειγμα, με τον ίδιο τρόπο και τι ίδιε αρχέ. Δεν κάνουμε τίποτα που να μην έχετε κάνει ήδη εσεί. Τώρα θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πολλά σημαντικά πράγματα, αλλά θέλω να επαναλάβω το εξή. Εμείς έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τη συζήτηση αυτή. Το νέο πλαίσιο που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνάντησε επικρίσεις στην προηγούμενη κυβέρνηση του Πρωθυπουργού κυρίου Τούσκ τότε. και μετά από διάφορες απόψεις και ε, γνωμοδοτήσεις ε, νομικών, ε, εμπειρογνωμόνων και άλλων, πού καταλήξαμε. Προτάθηκε ένα νέο πλαίσιο, το οποίο όμως ήταν απαράδεκτο για την Πολωνία. Έχω την αίσθηση ότι αδικούμεθα. Πάντως ήρθα εδώ, όπως βλέπετε, διότι θεωρώ ότι είναι καθήκον μου προς τη χώρα μου, προς την κυβέρνησή μου και το κοινοβούλιο μου, προς την Πολωνία πριν απ' όλα, της οποίας έχω την τιμή να είμαι ηγέτης, αλλά και από σεβασμό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να έρθω εδώ να σας εξηγήσω με λεπτομέρειες για το τι γίνεται στη χώρα μου. Αυτό είναι απαραίτητο. Απαραίτητο και για τη χώρα μου και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά όργανα. Πρόεδρος, τώρα λοιπόν ε, θα ακολουθήσουν οι επόμενοι μιλητές ε, που θα κλείσουν και τη συζήτηση θα έχουν ένα λεπτό χρόνο στη διάθεσή τους. Και πρώτα απ' όλα δίνω το λόγο στον κύριο Κόρμπιν Μίκε. Κύριε Πρόεδρε, άκουσα ότι ο κύριος Γκονζάλης Πόνς είπε ότι στην Ευρώπη υπάρχει μόνο το βασίλειο της δικαιοσύνης, ότι γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα, δημοκρατία και κράτος δικαίου. Πολλές φορές όμως ε, δυστυχώς είναι κανείς αναγκασμένος να επιλέξει μεταξύ των δύο. Όπως συμβαίνει συχνά στο Κοινοβούλιο, ε, ο ένας εκ των δύο κερδίζει και όσον αφορά το συνταγματικό δικαστήριο νομίζω ότι ε, ενημερωθήκαμε από την Πρωθυπουργό. Εγώ είμαι υπέρ της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, όμως η προηγούμενη κυβέρνηση σε αυτό το συνταγματικό δικαστήριο, στην περίπτωση αυτού, εξέτασε κατά πόσον ε, είναι συνταγματικά προβλέψιμο και θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι κάτι, ένα μόρφωμα το οποίο θα πρέπει να διαλυθεί. Äh, λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Μαρούζικ, ε, εκ του κόμματος της Ελευθερίας. Κυρίες και κύριοι, για να εξετάσει κανείς την κατάσταση στην Πολωνία δεν είναι εδώ ο σωστός χώρος. Αυτά που συζητούνται εδώ ε, συζητούνται στην Πολωνία, στους πολωνικούς θεσμούς. Γι' αυτό λοιπόν ας ε, είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι και ας δείξουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην Ευρώπη. Υπάρχουν πολλές ε, δυνάμεις που ήρθαν και έφυγαν, οι Ρωμαίοι, οι Σοβιετικένες και όλοι έφυγαν. Αλλά ακόμα κι αν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαλυθεί, θα εξακολουθεί να υπάρχει η Ευρώπη γιατί υπάρχουν πολλά κράτη που επιθυμούν το ίδιο, την ελευθερία και τη δικαιοσύνη. Γι' αυτό λοιπόν ας αφήσουμε αυτή τη συζήτηση, ας έχουμε πάντα κατά νου την Ευρώπη και να σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε για να μην εμπλεκόμαστε με αυτό που κάνουν όλοι οι άλλοι. Ας αφήσουμε όλους να ζουν με τον τρόπο που επιθυμούν. Ας αφήσουμε την Ευρώπη να είναι ελεύθερη, ας πιστέψουμε στην Ευρώπη. Και επιτρέψτε μου να προσθέσω και κάτι άλλο, γιατί από ό,τι φαίνεται έχω ακόμα χρόνο. Θέλω να σας πω, χαίρομαι πάρα πολύ για το γεγονός ότι αυτή η συζήτηση οδήγησε ε, στο να κληθεί κανείς να επιδείξει κοινό νου. Να παρουσιάσει τις ε, αντεγκλήσεις, τις ε, διαφωνίες κάτω από αυτό το πρίσμα, από το πρίσμα της λογικής του κοινού νου και νομίζω ότι τώρα πλέον ε, θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα πραγματικά προβλήματα της Ευρώπης. Και νομίζω ότι τότε θα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι λαοί που θα προωθηθούν και εξελιχθούν περαιτέρω. Εκ μέρους ε, της ε, EFDD, ο κύριος Ιβασκίβιτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Πρωθυπουργέ. Εγώ εκφράζω την αντιπολίτευση θα ήθελα να πω ότι η κοινοβουλευτική δημοκρατία λειτουργεί εγώ. Θα επιβεβαιώσω αυτό που είπαν οι δύο προηγούμενοι ομιλητές, ότι η συζήτηση αφορά τα σύνορα των αρμοδιοτήτων, τα όρια των αρμοδιοτήτων των θεσμικών οργάνων, τα οποία διευρύνονται όλο και περισσότερο, όλο και περισσότερες αρμοδιότητες προστίθενται, χωρίς καμία ουσιαστική δικαιολογία, χωρίς καμία ουσιαστική τεκμηρίωση. Οι κυβερνήσεις μόνες τους αποφασίζουν. Λοιπόν δεν θα πρέπει να υπάρχουν παρεμβάσεις στα εσωτερικά θέματα των χωρών. Ε, οι συμβουλές των Βέλγων πολιτικών ή των Ολλανδών πολιτικών αυτά να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας. Έχετε το πρόβλημα των μεταναστών που καταστρέφουν τις κοινωνίες σας, τους πολιτισμούς σας και δημιουργούν προβλήματα στις γυναίκες σας. Λοιπόν, Πρωθυπουργέ, συγχαρητήρια για αυτά που είπατε σήμερα. Νομίζω ότι το μέλλον της Πολωνίας είναι αποκλειστικά στα χέρια των Πολωνών, σε κανέναν άλλο. Από τους Πρασίνους, η κυρία Χάρς, παρακαλώ. Κυρία Πρωθυπουργέ, με πολλούς Πολωνούς συναδέλφους το το ε, χειμώνα του 2013 και του 2014 ήμασταν στο Euromaidan στο Κίεβο και μεταξύ αυτών και πολλούς δικούς σας συναδέλφους από το κόμμα σας οι οποίοι αγωνίστηκαν στεναρά για το κράτος δικαίου και για το δρόμο της Ουκρανίας προς τη Δύση και οπωσδήποτε κατά ε, ε της αυταρχικής επίδρασης του Κρεμλίνου και της οπισθοδρομικής και του κυρίου Πούτιν, όχι μόνο στην Ουκρανία και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να σας πω κάτι που με πονάει ειλικρινά στην αντίδρασή σας σε αυτή τη συζήτηση, ότι εσείς χειροκροτείτε βουλευτές οι οποίοι επιθετικά ζητούν την καταστροφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή και χρηματοδοτούνται γι' αυτό το λόγο από τον πρόεδρο Πούτιν. Αυτό παρακαλώ να το σκεφτείτε. Τι συμμαχίες κάνετε και να το ε, συζητήσετε και στην Πολωνία και αυτό. Γενικότερα τώρα θα ήθελα να πω κάποια πράγματα για τη συζήτηση. Πιστεύω ότι και πάλι έχουμε περιέλθει σε ένα σημείο που θα πρέπει να καταλάβουμε ότι Υπάρχουν και δυσάρεστες συζητήσεις για τους κανόνες του κράτους δικαίου, για τους δημοκρατικούς κανόνες, πράγματα τα οποία δεν ε, τηρούνται ενιαία ε, και δεν είναι ενιαία νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συζητήσεις που θα πρέπει επιγόντως να κάνουμε και την παραθέσεις. Γιατί πίσω από τη συζήτηση για το κράτος δικαίου στην Πολωνία υποβόσκει και αυτή η συζήτηση ε, τι μας κρατάει ενωμένους και γιατί δεν έχουμε καταφέρει να το ορίσουμε θετικά. Τι εστί η ευρωπαϊκή μας ταυτότητα. Γιατί έχουμε αυτές τις φυγόκεντρες τάσεις τώρα και μετά τις εκλογές και κρατών και λαών. Αυτό θα πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Πολωνία. Διότι εγώ ε, γνώρισα πολύ καλά την κοινωνία των πολιτών και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην πολωνική κοινωνία ότι δεν θα επιτρέψει η χώρα αυτή να κυβερνηθεί και πάλι με αυταρχικό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Τσίμερ από την ε, Νοτιοκία Ιστερά. Αξιότιμη κυρία Πρωθυπουργέ, ξέρετε όλη αυτή την ώρα σκέφτομαι γιατί αισθάνομαι ότι τελικά δεν ελέγχθησαν τα πράγματα με το όνομά τους. Και όπως και η Ρεμπέκα Χάρμς ε, και εγώ πρέπει να σας πω ότι με ενόχλησε ιδιαίτερα το ότι όταν έγινε λόγος για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κάποιοι από τους βουλευτές ε, είπαν ότι πρέπει να καταστραφεί, να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώς και εσείς θα συμφωνήσετε. Αυτό δεν ταιριάζει με αυτά που μας είπατε προηγουμένως. Εσείς διακηρύξατε ότι είσαστε Ευρωπαία, ότι είσαστε υπέρ της Ευρώπης και εσείς και το κόμμα σας είσαστε σε αυτή την ατραπό αλλά ξέρετε, αυτό που χρειαζόμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πτόντι, μία διόρθωση, μία σε βάθο μεταρρύθμιση. Αυτά που χρειαζόμαστε είναι να επανέλθει η Ευρωπαϊκή Ένωση στη βάση των αρχών της. Οι πολίτες να αισθάνονται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κάτι που τους προσφέρει υπεραξία, είναι κάτι που θέλουν να υπερασπιστούν, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η εναλλακτική εναλλακτική λύση στις σύγκρουσεις, στι εθνικές συγκρούσεις που βιώσαμε κατά το παρελθόν. Όλοι μας μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και γι' αυτό λοιπόν εγώ ήλπιζα ότι θα μας ε, δώσετε ένα μήνυμα ότι κατανοείτε πολύ καλά ότι η Πολωνία θα πρέπει να είναι η γέφυρα και είναι η γέφυρα ανάμεσα στην Ανατολή και τη Δύση. Αρκετοί ευρωβουλευτέ γνωρίζουν πολύ καλά τα προβλήματα στι ε, χώρε τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ότι υπάρχουν ακόμα πολλά που πρέπει να αναδιαταχθούν, αλλά ακριβώ εκεί αυτή είναι η δική σας η αρμοδιότητα και σας παρακαλώ να μην αποσύρεστε, να μην συγχαίρετε και χειροκροτείτε αυτούς τους κυρίους που ανέφερα προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι προσφέρετε οποιαδήποτε υπηρεσία στην Πολωνία με αυτόν τον τρόπο. Ο κύριος Φερχόφστατ. Θα πρέπει να σας πω ότι μετά από λίγε εβδομάδες χρησιμοποιείτε όλα τα τεχνάσματα και τα κόλπα των πρωθυπουργών. Μαθαίνετε πολύ γρήγορα. Είπατε ότι ήρθα να απαντήσω στι ερωτήσει σας. Ε, ακούσαμε τα σχόλια για το τι συμβαίνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ και άλλοι περιέγραψαν το πρόβλημα και δεν απαντήσατε. Και ποιο είναι το πρόβλημα με την αλλαγή στο συνταγματικό δικαστήριο. Επιτρέψτε μου να το εξηγήσω και πάλι. Μήπω θα διερμηνία, ξέρω εγώ, προς τα πολωνικά. Το, το σύστημα είναι απλό. Εσεί διορίσατε τρει, πέντε συνολικά νέους δικαστές στο συνταγματικό δικαστήριο. Τρεις εκ των οποίων με τους νέους κανόνες έχουν δικαίωμα βέτο για τρία μέλη μπορούν να μπλοκάρουν οποιαδήποτε απόφαση στο συνταγματικό δικαστήριο του κόμματός σας, είναι δικοί σας ε, δικαστές. Αυτή είναι η κατάσταση, αυτό συνέβη και δεν απαντάτε γι' αυτό. Το θεωρείτε απολύτως φυσιολογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και το μόνο επιχείρημα που έχετε είναι το είπε και ο κύριος Λεγκούτκο ότι η πλατφόρμα έκανε λάθη. Γεγονό, έκανε λάθη η προηγούμενη κυβέρνηση. Αλλά εσεί κερδίσατε τι εκλογέ για να τα πάτε καλύτερα από την πλατφόρμα, όχι να κάνετε κι εσεί τα ίδια λάθη με την πλατφόρμα. Αυτή είναι η δημοκρατία και κάνετε ακριβώ τα ίδια. Μα λέτε ότι εντάξει κάνανε και αυτοί διάφορα πράγματα μονοκομματικό κράτο και τώρα έχει έρθει η δική μα ώρα να κάνουμε εμεί το δικό μα μονοκομματικό κράτο για τα επόμενα χρόνια γιατί ήρθαμε εμεί τα πράγματα. Και έχω να σα κάνω την εξή μοναδική ερώτηση και νομίζω τουλάχιστον σε αυτό μπορείτε να απαντήσετε ως Πρωθυπουργό. Εάν η Επιτροπή τη Βενετία γνωμοδοτήσει αρνητικά, τι θα κάνετε. Θα ακολουθήσετε αυτή τη γνωμοδότηση τη Επιτροπή Βενετία. Ευχαριστώ πολύ. Α, μήπω να απαντήσει αμέσω, η Πρωθυπουργό. Καλά, ο κύριο Λεγκούτκο έχει το λόγο από τους συντηρητικούς. Ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε δύο σημαντικούς εχθρούς. Η άγνοια είναι ο πρώτος και η προκατάληψη ο δεύτερος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταπολεμήσει κανείς την προκατάληψη όσα μέσα και να έχει στη διάθεσή του. Έχουμε ένα συνταγματικό δικαστήριο, 9 προς 6 τα μέλη, λέει ο μιλητής, Αυτό σημαίνει βέβαια ότι με τον τρόπο με τον οποίο έχει διαμαρφωθεί η σύνθεση του δικαστηρίου δεν μπορεί στην παρούσα φάση να παίρνει αποφάσεις. Είναι βέβαια μια προσπάθεια η οποία έχει γίνει από τον νομοθέτη για να συνθέσει ένα δίκαιο κοινοβούλιο και είναι σαφές ότι δεν επιτρέπεται σε πέντε δικαστές να παίρνει αφαίρετες αποφάσεις. Ένα τέτοιο δικαστήριο είναι καλύτερο δικαστήριο, ακόμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το νέο λοιπόν συνταγματικό πολωνικό δικαστήριο είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Αυτά για το δικαστήριο να έλθω μία στιγμή τώρα στα μέσα ενημέρωσης. Έχουμε καλύτερα μέσα ενημέρωσης ή χειρότερα. Έχουμε μία ενιαία ρητορική η οποία βγαίνει από τα μέσα ενημέρωσης. Όχι βέβαια. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφοροποιήσεις και τι γίνεται με τους δημοσιογράφους οι οποίοι απολύθησαν από όλα τα μέσα ενημέρωσης 7-8 χρόνια πριν. Τώρα προσλαμβάνονται εκ νέου. Ευχαριστώ. Πρωθυπουργέ, στη συζήτηση που μόλις τελείωσε είναι τρεις οι γραμμές κατά την άποψή μου ταυτοποιούμε σαφώς. Πρώτον, μια γενική αποτίμηση φόρου τιμής στο ρόλο που διαδραμάτισε η Πολωνία ε, στην υπεράσπιση της κυριαρχίας καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας. Αναγνώριση των όσων έκανε η Πολωνία για να επανέλθει η δημοκρατία στην Ευρώπη. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ανησυχία που πλανάτε σαφέστατα για τις αποφάσεις που λαμβάνει η δική σας κυβέρνηση για τα μίντια και το συνταγματικό δικαστήριο. Κοιτάξτε, οι πάντες αναγνώρισαν ότι έχετε την εκλογική νομιμοποίηση, την επαρκή ακριβώς για να ε, κάνετε το, εκλογικό, το κυβερνητικό σας πρόγραμμα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Απλώς η πλειοψηφία, το γεγονό ότι έχετε δημοκρατικά την πλειοψηφία και τη δεδηλωμένη δεν σημαίνει ότι θα απεμπολούνται οι δημοκρατικέ αρχέ και δεν θα προστατεύεται η πολυφωνία και η πολυφωνία ελέγχεται με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο προ την κυβέρνηση και με την ελευθερία του τύπου. Διάφοροι ομιλητέ εξέφρασαν, ε, μάλλον άρχισαν να λένε εγώ είμαι Πολωνός. Και μάλιστα μερικέ φορέ είναι και κακέ παρέε και προσέχετε τι φιλίε σα. Θα ήθελα όμως να επαναλάβω αυτή την έκφραση. Θα σας πω ότι και εγώ Πολάκος, Πολωνό, θεωρώ ότι είμαι. Αλλά από όλου τους Πολωνούς που πήγαν να ψηφίσουν και του 50% που πήγε και του 50% που δεν πήγε, γιατί οι μισοί δεν συμμετείχαν. Και επειδή δεν συμμετείχαν στις εκλογές δεν σημαίνει ότι έχασαν τα δικαιώματά τους και από όσου ψήφισαν το 38% που σας έδωσε την νομιμότητα για να ε, κυβερνάτε και το 62 που ψήφισαν διαφορετικά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκονσάλεθ Πόνς έχει το λόγο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρωθυπουργέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τον τόνο και για την παρουσία σας εδώ στη μακρά αυτή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα μου άρεσε αυτά τα ωραία που είπατε ε, για την Ευρώπη εδώ να τα ακολουθεί και το κόμμα σας στην Πολωνία. Και όταν έρχεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λέτε θαυμάσια λόγια για την Ευρώπη και θα ήθελα να τα λέει τα ίδια το κόμμα σας και στην Πολωνία. Δεν με καθησύχασε αυτό που είπατε ότι είναι πολιτικό όργανο το συνταγματικό δικαστήριο. Δεν υπάρχουν τέτοια όργανα. Τα συνταγματικά δικαστήρια είναι νομικά όργανα. Δεν έχει νόημα να είναι πολιτικά. Και καθόλου δεν με καθησύχασε καθόλου αυτό που είπατε ότι η κυβέρνηση εγγυάται την ε, αντικειμενικότητα των μέσων ενημέρωση. Όταν ακούω να λέει η κυβέρνηση ότι θα εγγυηθεί την ουδετερότητα του τύπου, είναι σαν να έχεις βάλει το λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Ο τελευταίος που θα πρέπει να ασχολείται με αυτά τα θέματα και την αντικειμενικότητα είναι η κυβέρνηση, αν θέλουμε να υπάρχει ελευθεροτυπία. Και επαναλαμβάνω αυτό που είπα προηγουμένως. Δεν πρόκειται για τον νόμο. Έχετε και νομιμοποίηση να αλλάξετε ό,τι θέλετε. Οι αξίες είναι το θέμα που δεν μπορεί κανείς να τους αλλάξει. Και δεν πρόκειται για την Πολωνία στο κάτω-κάτω. Πρόκειται για την πολωνική κυβέρνηση. Δεν μπορείτε να συγχαίρετε τη χώρα με το κράτος. Αυτό είναι από τα πιο επικίνδυνα πράγματα που μπορεί κάποιο να κάνει στην πολιτική. Δεν πρόκειται για την κυριαρχία. Πρόκειται για το κράτος δικαίου. Δεν πρόκειται για την πολιτική, πρόκειται για την ελευθερία. Όπως έλεγε και ο Μάνφρετ Βέμπερ, πρόκειται για την ενότητα και όχι για τη διχόνοια. Και τελειώνω, όπως και ο Ερίκη Γκερέρο, λέγοντας ότι Ορισμένοι που είναι πολύ κακέ παρέ δήλωσαν σήμερα Πολωνοί. Όλοι οι Ευρωπαίοι μπορούμε να δηλώσουμε Πολωνοί γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Και το επαναλαμβάνω, είμαστε υπερήφανοι που είμαστε Ευρωπαίοι και είμαστε και Πολωνοί. Μια που κερδίσατε λοιπόν τις εκλογές, παρακαλούμε να μας διευκολύνετε τη ζωή να είμαστε Πολωνοί. Ευχαριστώ κύριε Γκοζάλης. Παρακαλώ. Η Πρωθυπουργός. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Και... Λοιπόν, εμείς περιμένουμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας. Να σας θυμίσω όμως ότι η πολωνική κυβέρνηση από μόνη της ζήτησε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής αυτής και δεν χρειαζόμαστε την ενθάρρυνση ουδενός για να το κάνουμε. Νομίζω ότι θα είναι πιο εύκολο να έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο και να χρησιμοποιήσουμε επιχειρήματα για να μην κάνουμε τη συζήτηση αυτή αν είχαμε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής γιατί είμαι βεβαία ότι η Επιτροπή θα δείξει ότι η κατάσταση νομική για, για το, το συνταγματικό δικαστήριο το ανώτατο της Πολωνίας είναι μια πολύ ε, θα έλεγα κανονική νομικά κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν οι 10 δικαστές να μπλοκάρουν τους 15 δικαστές στις ακραίες καταστάσεις. Νομίζω ότι αυτά είναι επιχειρήματα γνωστά, θέλω να σας τα παρουσιάσω και πάλι, αν και θεωρώ ότι η συζήτηση την οποία οργανώσατε εδώ σήμερα είναι μια συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου. Είμαι όμως εδώ γιατί σέβομαι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, θεμητό είναι να θέλει να ασχοληθεί με το θέμα αυτό το οποίο μπορεί να θεωρεί προβληματικό. Δεν θα αναφερθώ σε κάποιες παρεμβάσεις τις οποίες θα θεωρήσω εκτός τόπου συγκεκριμένα. Έχω και εγώ ένα επίπεδο αξιοπρέπειας σαν πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που με το επιβάλλει αυτό. Εμείς δεν είμαστε εθνικιστές. Το κόμμα μου δεν είναι εθνικιστικό και μας προσβάλλει που χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο επιθετικό προσδιορισμό. Να επαναλάβω όμως το εξής. Η πολωνική κυβέρνηση εξελέγει με δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές από τον πολωνικό λαό να επαναλάβω ότι η πολωνική κυβέρνηση διαχειρίζεται την Πολωνία σήμερα γιατί έχει την εντολή του λαού. Δεν είναι λοιπόν κάτι εκτός, κάτι το διαφορετικό από τη χώρα. Απλά σεβόμεθα τους δημοκρατικούς κανόνες και εσείς το ίδιο κάνετε στις δική σας χώρες. Δεν θα βγω εγώ να πω δεν σέβομαι εγώ την κυβέρνηση της Ολλανδίας ή την κυβέρνηση της Ισπανίας. Όχι βέβαια, σέβομαι την Ολλανδία, σέβομαι την Ισπανία και σέβομαι και τις κυβερνήσεις τους. Προφανώς ο καθένας μπορεί να έχει τις δικές του απόψεις και αυτή η διαφοροποίηση είναι τα θεμέλια της Ευρώπης. Έχουμε διαφορές. Πολλές φορές διαφωνούμε, αλλά συζητάμε τις διαφορές μας, συζητάμε τις διαφωνίες μας, και αυτό συνιστά την προστιθέμενη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πολωνία και τους Πολωνούς πολίτες. Για πάρα πολλά χρόνια εμείς στην Πολωνία δεν είχαμε την δυνατότητα να συζητάμε τα θέματα ελεύθερα. Μιλάτε για τη δικαιοσύνη, μιλάτε για την ισότητα και καλά κάνετε που τα συζητάτε τα θέματα αυτά. Καλό είναι να ασχολείστε επίσης και με τα προβλήματα της οικονομίας στην Πολωνία, τα προβλήματα των πολωνικών φτωχότερων περιφερειών, της Σιλεσίας. Εγώ σέβομαι τα θέματα τα οποία θέσατε και για τη Σιλεσία. Είμαι από την περιοχή πολύ κοντά στην Σιλεσία, είναι μια πανέμορφη χώρα, μια πανέμορφη περιοχή, συγγνώμη, η οποία χρειάζεται οικονομική βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Οι κάτοικοι της Σιλεσίας μου λένε συνέχεια θα μας βοηθήσει επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας. Κατανοεί η Ευρώπη ότι έχουμε ανάγκη τη βοήθειά της ή θα μας αμφίσει να βουλιάξουμε όπως τα πολωνικά ναυπηγεία. Λοιπόν, αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία τίθενται από τους Σιλεσιανούς. Αυτά είναι τα ερωτήματα τα οποία τίθενται από τους Πολωνούς. Οι Πολωνοί πρέπει να νιώσουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πλάι τους όταν τους έχει ανάγκη. Γι' αυτό είμαι εδώ σήμερα, γιατί πιστεύω στην Ευρώπη. Γιατί πιστεύω ότι η κοινωνία των πολιτών στην οποία επανειλημμένα αναφερθήκατε συνεργάζεται με την κυβέρνησή μας και εμείς είμαστε διαθέσιμοι να συνεργαστούμε μαζί της. Γιατί τα θέματα αυτά θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουμε ένα συγκεκριμένο αρμόδιο για τα θέματα της κοινωνίας των πολιτών. Να θυμίσω ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν τέτοιου είδους θέσεις. Εγώ έχω ασχοληθεί προσωπικά με την κοινωνία των πολιτών και έχουμε τρομερά παραδείγματα στην ιστορία μας όπως το κίνημα της αλληλεγγύης, θέματα που άπτονται της κοινωνίας των πολιτών που αποτελούν σήμερα τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζουμε την κοινή Ευρώπη, την Ευρώπη των ανεξαρτήτων χωρών. Αυτό κάνουμε, αυτό θα κάνουμε και με τη βούληση του πολωνικού λαού εμείς θα διαχειριστούμε τη χώρα με τον τρόπο με τον οποίο η Πολωνία επιθυμεί. Η Πολωνία σέβεται τον νόμο, η Πολωνία σέβεται το Σύνταγμα και σέβεται και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω, είμαι Ευρωπαία, είμαι υπερήφανη που είμαι Ευρωπαία, αλλά πριν είμαι Ευρωπαία είμαι Πολωνή. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Πρωθυπουργέ. Διακόπτει ο πρόεδρος ή διακόπτεται. Δυστυχώς η συζήτηση με τον κύριο Φεχόφτσατ γίνεται εκτός μικροφώνου και εμείς δεν ακούμε τίποτα. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται υπάρχει κάποιο πρόβλημα μετάφρασης γιατί η πρωθυπουργή υπουργό μίλησε πολωνικά. Εγώ παρακολούθησα τη διερμηνία στα αγγλικά, αλλά δεν κατάλαβα. Ε, να το ξαναπούμε. Είπατε ότι θα <laughs> δεχθείτε αυτά που θα αποφανθεί η ε, πιτροπή της ε, Βενετίας ή όχι. αν πείτε ένα σκέτο ναι ή όχι, θα το καταλάβω και στα πολωνικά να το πείτε. Ναι ή όχι, πέστε μας. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διερμηνίας, σας διαβεβαιώ. Ε, κατανοώ ότι θυμώνετε γιατί ε, θα θέλατε να ακούσετε κάτι διαφορετικό αλλά εγώ επιτρέψτε μου να σας πω ότι ήρθα εδώ, διένυσα μια απόσταση πάρα πολλών χιλιόμετρων για να διαλύσω οποιασδήποτε αμφιβολίες και δεν έχω κανένα πρόβλημα θα ήθελα λοιπόν να κατανοήσετε ότι πρέπει η μία πλευρά να ακούει την άλλη. Και εκείνο το οποίο οφείλουμε να κάνουμε είναι να θέλουμε να ακούσουμε. Γι' αυτό λοιπόν ας μιλήσουμε για γεγονότα και όχι για προκαταλήψεις. Ε, το θέμα δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί. Περιμένουμε ακόμα τη γνωμοδότηση και μόλις δημοσιευτεί η γνωμοδότηση θα την αναλύσουμε ενδελεχώς, ενδελεχέστατα μάλιστα. Ευχαριστώ κυρία Πρωθυπουργέ. Ο κύριος Κούντας έχει το λόγο, ξέρω με το Συμβουλίο. Ναι, κοιτάξτε κύριε Φερχόστατ. Εντάξει, αυτή είναι η απάντηση. Είναι σκληρή για σας, το καταλαβαίνω, αλλά δουλέψτε το, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, Πρωθυπουργέ, αξιότιμα μέλη. Πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση, αλλά και πάρα πολύ ευαίσθητη φάνηκε ξεκάθαρα από ε, τη τελευταία συζήτηση τώρα. Πάντως ήταν πάρα πολύ σημαντική. Όλοι μας και όλοι σας μιλήσατε για τη σημασία του κράτους δικαίου ως θεμελιώδη λίθο της συνεργασίας μας. Με πάρα πολύ λίγες αλλά, ε, εξαιρέσεις, ελάχιστες αν υπήρχαν. Θετικά είναι αυτά. Αλλά όταν μιλούμε για κράτος δικαίου, από ό,τι φαίνεται, πολύ γρήγορα δεν είναι μόνο νομικό ζήτημα αλλά και πολιτικό. Και αυτό είναι κατανοητό κατά τα άλλα. Είναι ένα ζήτημα κυριαρχίας, ε, θεσμικής ισορροπίας ε, και κρισίμων ε, περιπτώσεων. Και γι' αυτό η συζήτηση για το κράτος δικαίου είναι γενός πολιτική και πάρα πολύ σημαντική να γίνεται εδώ στο Κοινοβούλιο. Νομίζω όλοι ξεκαθαρίσατε ότι θα πρέπει να μην υπάρχουν διπλά, ε, διπλές προδιαγραφές ε, και κανένας δεν είναι δακτυλοδικουκτούμενος. Όλοι μας ζούμε ένα πολύ δύσκολο διάστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει ο καθένας να κοιτάξει τα θεμέλια του κράτους δικαίου στη χώρα του. Εγώ μιλώ εδώ εξ ονόματος του Συμβουλίου Υπουργών δεν έχουμε συνεδριάσει για αυτό το θέμα ακόμα, αλλά προσπαθώ να σας διαβεβαιώσω και ότι από πλευρά του Συμβουλίου είναι πολύ σημαντικό το θέμα του κράτους δικαίου και έχουμε συμφωνήσει για διάφορα θέματα. Το ένα έχει να κάνει με το νέο μηχανισμό που ίδρυσαν Συμβούλιο και Επιτροπή ένα αιτήσιο διάλογο για το κράτος δικαίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει και ένα αντίστοιχο πλαίσιο το Μάρτιο του 2014. Τώρα πρόκειται να τεθεί σε ισχύ αυτό ο μηχανισμό και έγινε και μια ερώτηση σε ποιο βαθμό θέλουμε ένα ενισχυμένη συνεργασία ή κάποιο άλλο μηχανισμό. Ακόμα δεν έχω δει ε, την έγκριση της πρότασης Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα το εξετάσουμε, θα το μελετήσουμε και είναι σημαντικό να αρχίσει το Κοινοβούλιο να ε, το επεξεργάζεται σε πλήρη σεβασμό και διάλογο όλων των ενδιαφερόμενων μερών και σε συνεργασία όλων των θεσμικών οργάνων. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν θα έλεγα εξ της Προεδρίας ότι όπως γνωρίζετε είμαστε προσιλωμένοι στο σεβασμό των θεμελιωδών και βασικών ε, αρχών της Ένωσης και αξιών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα αναλύει τα γεγονότα, είναι σε διαρκή διάλογο με την πολωνική κυβέρνηση και ε, είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος ε, της παρακολούθησης αυτών των θεμάτων παντού στην Ένωση, ιδιαίτερα επειδή είναι θεματοφύλακας των ε, συνθήκων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ξέρετε ποια είναι η θέση της Προεδρίας, ποια είναι η θέση του Συμβουλίου και είχατε την ευκαιρία σήμερα να συζητήσετε με την Πολωνή Πρωθυπουργό και ήταν και ίδια που θέλησε να έρθει εδώ να ακούσει τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας. Εγώ τι αποκόμισα από τη συζήτηση αυτή, από το πνεύμα που πριτάνευσε. Ότι καμιά φορά είναι ευαίσθητα αυτά τα θέματα, αλλά πρώτα απ' όλα χρειάζεται διάλογος. Όλοι συμφωνούν ότι χρειάζεται σοβαρός διάλογος. Δεύτερον, από όλε τι πλευρέ το άκουσα επίση ότι πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί, να κοιτάμε τα αντικειμενικά γεγονότα με τρόπο νυφάλαιο και σε πνεύμα συνεργασίας που είπε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ήταν σημαντικό που αναφέρθηκε η Επιτροπή της Βενετίας εδώ. Και να είστε βέβαιοι ότι η Προεδρία θα το παρακολουθήσει όσο γίνεται πιο σκενά και θα αγωνιστεί από κοινού. Έχουμε διάφορα μέσα στη διάθεσή μας, άρθρα, συζητήσεις, επιστολές και το κράτος δικαίου θα συνεχίζει να ανθεί και να αναπτύσσεται στην Ευρώπη. Διότι Μόνο σε μια τέτοια ε, κατάσταση μπορεί να αναπτυχθεί μια παλόμενη κοινωνία. Και από πολιτική σκοπιά το κράτος δικαίου είναι ε, και άχρωμο, δεν κοιτάει χρώματα και κομματικές τοποθετήσεις. Είναι, έχει χρωματοψία μάλλον. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Πρώτο ο κύριο Σόιτιγκερ. Κυρία Πρωθυπουργέ, κυρίε και κύριοι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα μέσα ενημέρωσης ε, έχουν ε, μια δική του σημασία. Η ανεξαρτησία των μέσων ενημέρωσης είναι ένα πολύτιμο αγαθό. Το ίδιο ισχύει και για την πολυμορφία στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Ε, γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν εφόσον υπάρχουν καταγγελίες, έχει όχι μόνο το δικαίωμα, αλλά και την υποχρέωση να ελέγχει κατά πόσον πράγματι στην Ευρώπη υπάρχει κίνδυνος για την ανεξαρτησία και την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Και αυτό ακριβώς καλούμεθα να κάνουμε. Τίποτα παραπάνω, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Στο νέο νόμο περί μέσων ενημέρωσης ε, στην Πολωνία προβλέπονται τρία όργανα το ε, Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο, της ΤΕΦΑΟΠΕ και της ΕΦΑΟΠΕ, δηλαδή της δημόσιας ε, τηλεόρασης και του δημόσιου ραδιοφώνου της Πολωνίας. Πρόκειται για το Εποπτικό Συμβούλιο και για τα δύο όργανα και πρόκειται και για τον, ας τον πούμε, διαμεσολαβητή των μέσων ενημέρωση. Μέχρι τώρα λοιπόν το Εποπτικό Συμβούλιο ε, συνετίθετο από 7 μέλη. Ως εξής, πρώτον, ένας, μία πρόταση από τον Υπουργό Πολιτισμό, μία πρόταση από την, ε, τον ε, Πρωθυπουργό, άρα δύο ή τρεις και οι υπόλοιποι από τον διαμεσολαβητή από τη ρυθμιστική αρχή. Αυτό που είναι καινούριο και αποφασίστηκε στο τέλος του έτους, το από 7 πάμε σε 3 μέλη και οι 7 αποφασίζονται όλοι από τον Υπουργό Επικρατείας. Το δεύτερο που θέλω να πω όσον αφορά το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο στο μέλλον χωρίς ε, καμία αιτιολογία και ανα πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να συγκληθεί και να παυτεί. Αυτή λοιπόν την απόφαση τη λαμβάνει και πάλι το Εποπτικό Συμβούλιο, το οποίο όπως σας είπα ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από τον Υπουργό Επικρατείας. Στο καταστατικό της δημόσιας τηλεόρασης και του δημόσιου ραδιοφώνου προβλέπεται χωρίς τον ε, ε, τη ρυθμιστική αρχή και χωρίς το κοινοβούλιο να μπορούν να υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Εμείς λοιπόν προβληματιζόμαστε γιατί ε, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι τα κόμματα αλλά μόνο η κυβέρνηση που μπορεί να περικόψει την ανεξαρτησία του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης. Αυτό είναι το ερώτημα που τίθεται και ε, το εξετάζουμε ε, και είμαστε ευγνώμονες που η κυβέρνηση μας είπε ότι θα υπάρξει διάλογος. Εμείς ε, θέλουμε να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος μέσα από το νόμο περί μέσων ενημέρωσης που θα συζητηθεί Φεβρουάριο ή Μάρτιο. Θέλουμε να πιστεύουμε τότε θα υπάρχει η ευκαιρία για τη συνέχεια του διαλόγου και θα ήταν βέβαια πολύ καλύτερα αν τα θέματα περί ε, εφταξίας και κράτους δικαίου να μην εξετάζονται αναδρομικά αλλά την κατάλληλη, την τρέχουσα στιγμή ε, πριν από την λήψη απόφασης να γίνεται συζήτηση με τα αρμόδια όργανα. Πολύ ωραία. Για να κλείσω το θέμα, το λόγο έχει ο κύριος Τίμερμανς, αντιπρόεδρος της Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε και αγαπητά μέλη. Υπάρχουν πάρα πολλά επί των οποίων θα μπορούσε κανείς να τοποθετηθεί σήμερα, αλλά λόγω της προκεχωρημένης ώρας θα είμαι πολύ σύντομος. Τρία πράγματα. Πρώτον, έχοντας ακούσει όλα αυτά για την κυριαρχία, εγώ θεωρώ ότι η Πολωνία τώρα είναι περισσότερο κυρίαρχη, είναι περισσότερο αφεντικό ας το πούμε της ε, μοίρας της, πολύ περισσότερο τώρα από ό,τι ήταν πριν, πριν γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα έχει ενώσει την κυριαρχία της με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για πρώτη φορά σύνορα που δεν τα αμφισβητούν οι γείτονε. Ε, κυρία Πρωθυπουργέ, αυτή είναι η πραγματική κυριαρχία. Αυτό είναι το πραγματικό επίτευγμα όλων των ευρωπαϊκών κρατών, πόσο μάλλον της Πολωνίας. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι όλα τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν διακηρύξει τη βούλησή τους ε, και ε, έχει επιβεβαιωθεί αυτό από τα κοινοβούλια. Άρα δηλαδή έχουν τη δέσμευση να διαφυλάσσουν το κράτος δικαίου. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να επιτρέπουν και να κρίνονται από το δικαστήριο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο ε, Λουξεμβούργο να κρίνονται από την Κομισιόν και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν θέλετε ε, να αμφισβητούνται και από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δηλαδή οποτεδήποτε τίθεται θέμα ε, κράτους δικαίου δεν μπορεί κανείς να κρύβεται πίσω από την εθνική κυριαρχία. Δεν γίνεται αυτό γιατί έχετε υπογράψει και λέτε ε, με την υπογραφή σας ότι τέτοιου είδους θέματα συζητούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κύριος Ντεκούτο του αρέσουν πάρα πολύ τα γεγονότα. Μα αυτά που σας λένε γεγονότα και να σας πω και άλλα σχετικά παρεπιπτόντω, και εντεγκουτικό. Πράγματι, έχετε απόλυτα δίκιο ότι μπορεί κανεί να έχει την άποψή του, αλλά ξέρετε δεν μπορεί κανεί να έχει τα δικά του τα στοιχεία. Αυτό δεν γίνεται. Θα θίξω λοιπόν κάποια θέματα. Ε, κυρία Πρωθυπουργέ, εμεί δεν έχουμε καμία αντίρρηση ε, όσον αφορά την αρχή ότι η σύνθεση του σταγματικού δικαστηρίου θα πρέπει να είναι ισορροπημένη. Συμφωνούμε επίση ότι το σταγματικό δίκαιο θα πρέπει να γίνεται σεβαστό στην Πολωνία. Εκείνο όμω που μας ανησυχεί είναι ότι το συνταγματικό δικαστήριο έχει ερμηνεύσει και εφαρμόσει νόμους ε, και οι αποφάσεις του όμως ε, έχουν γίνει μερικώς μόνο αποδεκτές από εσάς. Εγώ δεν αναφέρομαι στην απόφαση της 30ης ε, Δεκεμβρίου που το δικαστήριο λέει ότι το παλιό, η παλιά κυβέρνηση είχε διορίσει πολλούς δικαστές. Εγώ αναφέρομαι στην απόφαση της 9ης Δεκεμβρίου όπου το συνταγματικό δικαστήριο ενέκρινε ένα νόμο που καταργεί όλους τους τους παλαιότερους διορισμούς συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είχαν γίνει με την έγκριση του Κοινοβουλίου. Άρα δηλαδή στο διάλογο όμως που θα συνεχιστεί παρακαλώ να τοποθετηθείτε επ' αυτού. Και κάτι άλλο, εάν σας αρέσει και συμφωνεί τόσο πολύ με την ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, της Βενετίας γιατί τη ζητήσατε όπως μας το είπατε και σήμερα, τότε γιατί δεν περιμένετε να εφαρμόζονται οι νόμοι μέχρι να τοποθετηθεί και η Επιτροπή της Βενετίας. Γιατί τώρα έχετε προτρέξει. Άρα δηλαδή η απόφαση ή η γνωμοδότηση της Επιτροπής Βενετίας θα έρθει εκ των υστέρων. Και παραμένει το ερώτημα πώς θα λύσει τα θέματα αυτά η Πολωνία. Γιατί μόνο αν λυθεί το θέμα της σύνθεσης του δικαστηρίου, μόνο τότε το δικαστήριο του συνταγματικού της Πολωνίας θα μπορεί και πάλι να παίξει το ρόλο του που είναι θεματοφύλακας του κράτους δικαίου στην Πολωνία. Επίσης να πω το κράτος δικαίου και ιδιαίτερα ο διαχωρισμός των εξουσιών, η διάκριση μάλλον των εξουσιών είναι κάτι που μας απασχολεί όλους μας. Μέσα από αυτή την επώδυνη ευρωπαϊκή ιστορία έχουμε μάθει ότι χρειαζόμαστε αυτό το τρίγωνο. Δημοκρατία, σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα και σεβασμό για το κράτος δικαίου. Αυτό το τρίγωνο δεν μπορεί να ισορροπεί αν ε, κάποια πλευρά παραπέει. Δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τη δημοκρατία ως επιχείρημα έναντι του κράτους δικαίου ούτε τη δημοκρατία ως επιχείρημα κατά του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Με πόνο και κόπο το μάθαμε αυτό και η Πολωνία ανέκαθεν η πάντα ήταν το μεγαλύτερο θύμα αυτής της οδυνηρής ιστορίας. Τώρα λοιπόν έχουμε μια ελεύθερη, ανεξάρτητη Πολωνία, όχι ανεξάρτητα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακριβώς λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό να διατηρήσουμε τον επικοδομητικό διάλογο με την πολωνική κυβέρνηση, γιατί είμαι πεπισμένος ότι αυτά τα θέματα μπορούμε να τα λύσουμε σεβόμενοι τους κανόνες τους οποίους έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει να σας παρακαλέσω να ολοκληρώσετε. Και εσείς, ε, κυρία Πρωθυπουργέ, ζητήσατε πάλι το λόγο, κύριε Σίτλο. Προφανώς είστε προσκεκλημένοι ε, ε, και δεν μπορώ, ούτε θέλω να σας αρνηθώ αυτό το δικαίωμα. Θα πρέπει να σας πω όμως ότι θα ξαναρχίσει η συζήτηση αν ξαναπάρετε το λόγο. Και σύμφωνα με τον κανονισμό δεν μπορώ να κάνω κάτι τέτοιο, διότι με τις ε, δηλώσεις του κυρίου Τίμερμαν ολοκληρώθηκε η συζήτηση. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτά που θα μας πείτε θα έχει χαρακτήρα τώρα ενημερωτικό γιατί δεν μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω συζήτηση, να μην είναι τρίτο ε, τριτολογία, αλλιώς θα πρέπει να πάρουν το λόγο και οι συνάδελφοι. Παρακαλώ, Πρωθυπουργέ, έχετε το λόγο. Ε, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, για την ευγένειά σας που μου δώσατε τον λόγο εκ νέου. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για μια σημαντική συζήτηση και για την χώρα μου αλλά και για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύω. Σας ευχαριστώ πολύ και υπογραμμίζω ξανά ότι η Πολωνία είναι μια δημοκρατία, είναι μια χώρα κράτος δικαίου που σέβεται το συνταγματικό της χάρτη, που σέβεται τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας, τις δηλώσεις σας, τα σχόλιά σας. Ελπίζω ότι οι πληροφορίες τις οποίες σας έδωσα θα σας επιτρέψουν να διαμορφώσετε μια καλύτερη εικόνα. Από δικής μας πλευράς να αναφερθώ σε αυτό το οποίο ζήτησε ο Επίτροπος γιατί να μην περιμένουμε την γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας. Κοιτάξτε, εμείς υιοθετήσαμε ε, μια νομοθετική ρύθμιση για το συνταγματικό δικαστήριο που με τη σειρά του ε, είχε, ε, αν θέλετε, τροπολογήσει μια προηγούμενη νομοθετική ρύθμιση η οποία παρουσίαζε θέματα σύμφωνα με το ίδιο το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Κοιτάξτε, δεν περιμέναμε, όπως και εσείς δεν περιμένατε πριν κάνετε τα σχόλιά σας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως και το Κοινοβούλιο δεν περίμενε πριν οργανώσει την συγκεκριμένη αυτή συζήτηση. Πάντως, τέτοιου είδους συζητήσεις ε, μας ε, φέρνει σε επαφή και επικοινωνούμε καλύτερα. Πρωθυπουργέ, Πρωθυπουργέ, Πρωθυπουργέ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ihre Intervention για την παρέμβασή σας και σας ευχαριστώ επίσης και για τις ευχαριστήσεις που απευθύνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα και προσωπικά να σας ευχαριστήσω, Πρωθυπουργέ, το γεγονός ότι ήρθατε εδώ ε, και ε, συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση και σταθήκατε στο Κοινοβούλιο και αυτό σας ε, διαφοροποιεί πάρα πολύ από εκείνους που σας χειροκροτούν, που λέγουν ότι δεν έχει καμιά δουλειά εδώ η συζήτηση. με πολύ ευεργετικό τρόπο διαφέρεται από τους υπολοιπούς.